Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, να ξεκινήσουμε. Θα έχουμε την παρουσίαση μιας μελέτης για τα αυτοοδηγούμενα οχήματα, το μέλλον της κυκλοφορίας οχημάτων και το μέλλον ε, το, της οδικής κυκλοφορίας στην εποχή των νέων τεχνολογιών. Οπότε συνδυάζεται με τη συνάντηση που είχαμε στο Άμστερνταμ. Χαιρετίζω τους προσκεκλημένους μας που θα μας παρουσιάσουν ε, τις θέσεις τους. Πρώτα απ' όλα βέβαια θα μας παρουσιάσουν την έρευνα για τα αυτοοδηγούμενα οχήματα, το μέλλον της οδικής κυκλοφορίας η κυρία Φριζόνη λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μας δίνει την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της μελέτης μας. Ήταν βέβαια δύσκολο το καθήκον μας. Πρώτα απ' όλα χρησιμοποιήσαμε τους ορισμούς για τα αυτόνομα οχήματα και μία παρουσίαση των ε, προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Ορισμένα δύσκολα ερωτήματα ήταν να καθορίσουμε το μέλλον αυτών των τεχνολογιών και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις για τους χρήστες ε, της οδικής κυκλοφορίας και την κοινωνία γενικότερα και καθώς ε, και μερικές συστάσεις για το τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το τομέα. Η μελέτη μας ασχολήθηκε κυρίως με την αυτοματοποίηση των οχημάτων. Όποιοι ξέρουν το θέμα και είναι πολύ σήμερα, ξέρετε ότι υπάρχει μια σαφής διάκριση μεταξύ της αυτοματοποίησης των οχημάτων και της συνδεσιμότητας των οχημάτων. Αλλά όταν συζητάμε τις ενδεχόμενες επιπτώσεις για να καθορίσουμε το μέλλον ε, των μεταφορών. Αυτοί οι δύο ορισμοί, σύνδεση των οχημάτων και αυτοματοποίηση των οχημάτων, δηλαδή πώς συνεργάζονται μεταξύ τους τα οχήματα, αυτή είναι η σύνδεση, πώς ε, ε, επικοινωνούν με την υποδομή μεταφορών ή με τα smartphone, αυτά συνδυάζονται σε πολλές περιπτώσεις. Ιδιαίτερα αν θέλουμε να δούμε τις ενδεχόμενες επιπτώσεις. Εδώ υπάρχει ε, μία δήλωση από την, ε, μία παράθεση από την ε, διακήρυξη του Άμστανταμ για να θέσουμε το πλαίσιο. Εδώ βλέπετε την ταξινόμηση που υπάρχει και για τα αυτοματοποιημένα οχήματα και για τη σύνδεση δηλαδή την πληροφορικοποίηση των οδικών μεταφορών. Στη μελέτη μας καθορίσαμε, εντοπίσαμε μάλλον, διάφορες τεχνολογίες που είναι υπό ανάπτυξη ή που ήδη είναι στην αγορά για τα διάφορα επίπεδα αυτοματοποίησης. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας ε, περιγράψω λεπτομερώς όλα αυτά, αλλά για να θέσουμε ένα πλαίσιο στη συζήτηση πρέπει να πούμε ότι η πλήρης αυτοματοποίηση είναι μόνο η κατάληξη μιας ολόκληρης διαδικασίας όπου θα περάσουμε από διάφορα επίπεδα αυτοματοποίηση. Βλέπετε εδώ στο κάτω μέρος τη διαφάνεια ότι υπάρχουν πέντε επίπεδα αυτοματοποίηση. και η πλήρως αυτόματη οδήγηση είναι μόνο το τελευταίο. Το άλλο σημείο που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι μεταξύ των επιπέδων 3 και 4 υπάρχει μια σαφής διαχωριστική γραμμή. Γιατί όλες οι τεχνολογίες που ήδη είναι υπό εξέλιξη ή ήδη σε χρήση βασίζονται στον οδηγό. Είναι γύρω από τον οδηγό, με κέντρο τον οδηγό. Οδηγό και αντρικέ για να βοηθήσουν τον οδηγό να αυξήσουν την άνεση και την ασφάλεια. Αλλά αν περάσουμε στα επίπεδα 4-5, τότε αλλάζει εντελώ ε, η προσέγγιση. Το όχημα ε, μπορεί να λειτουργήσει, θεωρητικά τουλάχιστον, αυτόματα, από μόνο του. Στη μελέτη μας Κάναμε μία αξιολόγηση των διαφόρων ε, τεστ. Πολλές γίνονται με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ένωση και κάναμε και μία επισκόπηση των διαφόρων ενδιαφερομένων. Πολλές διαφορετικές οργανώσεις και οργανισμοί και φορείς συμμετέχουν. Και εξετάζοντας τι συμβαίνει, στην Ένωση, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ιαπωνία, προσπαθήσαμε και να ταξινομήσουμε τι συμβαίνει και εντοπίσαμε τουλάχιστον για τα ΙΟΤΑΧΗ δύο προσεγγίσεις. Διαπιστώσαμε ότι οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες αλλά και άλλοι φορείς έχουν μια προσέγγιση που θα μπορούσαμε να την περιγράψουμε ως εξελικτική, όπου η αυτοματοποίηση των οχημάτων είναι μια σταδιακή διαδικασία. Και η πλήρως αυτόματη οδήγηση είναι μόνο, όπως είπα, η κατάληξη. Αντίθετα, άλλοι φορείς έχουν διαφορετική προσέγγιση, που θα μπορούσαμε να την πούμε επαναστατική οι πιο αξιόλογοι είναι μάλλον το Google. Αυτοί οι φορείς προσπαθούν να επιτύχουν απευθεία την πλήρως αυτόματη οδήγηση. δεν ενδιαφέρονται για τα χαμηλότερα επίπεδα αυτοματοποίησης. Λοιπόν, μέχρι εκεί εύκολα τα πράγματα. Τώρα, όταν προσπαθήσαμε να προβλέψουμε το μέλλον, συζητήσαμε με διάφορους ειδήμονες, ε, συζητήσαμε για διάφορα υλικά, για διάφορες προσεγγίσεις μάλλον. Δεν υπάρχει ενιαία άποψη για το τι θα γίνει στο μέλλον. Εμείς θεωρούμε ότι τα ΙΧ ή γενικότερα τα οχήματα με επιβάτες για να περάσουν από το 2 στο 4 δεν θέλουν πολύ χρόνο. Πολλές τεχνολογίες είναι ήδη ε, στην αγορά και πιο εκλεπτισμένες θα προκύψουν στα επόμενα 10-20 χρόνια πιο προωθημένες. Δεν περιμένουμε την πλήρη αυτοματοποίηση να προκύψει πολύ σύντομα. Πιστεύουμε ότι αργότερα θα προκύψει, ας πούμε, ίσως ε, περίπου σε 20 χρόνια. Ακόμη και αν κάποιες συγκεκριμένες εφαρμογές για συγκεκριμένες καταστάσεις θα μπορούσαν να εισαχθούν νωρίτερα. Αλλά για τα εμπορεύματα, α, και την ε, την αυτοκινητοπομπή φορτηγών, την πομπή. Θεωρούμε ότι και πάλι εδώ θα είναι σταδιακή η επίτευξη αυτού του στόχου. Θα δούμε ότι οι ευθύνες των οδηγών που θα κάθονται στο κουβούκλιο θα μειώνονται σταδιακά και αναμένουμε ότι η πλήρης αυτοματοποίηση είναι πιο μακροπρόθεσμη η προοπτική. Για τα αστικά όμως τώρα περιβάλλοντα και τις ε, συγκοινωνίες, τις δημόσιες μεταφορές, είναι κάπως διαφορετική η κατάσταση. Γιατί η ανάπτυξη πλήρως αυτοματοποιημένων οχημάτων σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, για παράδειγμα αεροδρόμια, εκθεσιακά κέντρα, συγκεκριμένε διαδρομέ, συγκεκριμένες περιοχέ, αυτό θα μπορούσε να συμβεί ακόμη ταχύτερα. Επίσης μελετήσαμε διάφορες άλλες επιπτώσεις. Βλέπω ότι λίγει ο χρόνος μου. Λοιπόν, τι επιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα οδική ασφάλεια. Όλοι γνωρίζουμε ότι 90% περίπου των ατυχημάτων ε, οφείλονται σε ανθρώπινο σφάλμα. Άρα πολύ, πολλά περιθώρια για την πληροφορική και την αυτοματοποίηση να βελτιώσουν εδώ την κατάσταση. Και γενικότερα η απόδοση από πλευράς ασφάλειας των αυτοματοποιημένων συστημάτων πρέπει ακόμη να αποδειχθεί. Ε, Εξετάσουμε εντελεχώς το θέμα αυτό. Τώρα, σε τι βαθμό η αυτοματοποίηση των οχημάτων θα βελτίωνε την ασφάλεια στους δρόμους. Θα είχε να κάνει με το ποσοστό συμμετοχή τους ε, ε, στο σύνολο των κυκλοφορούν των οχημάτων. Και αυτό θα είναι μια πιο μακροσκελής διαδικασία. Ε, εξετάσαμε και άλλα στοιχεία, για παράδειγμα εκπομπές και τέτοια περιμένουμε ότι θα μειωθεί το κοινωνικό κόστος των ε, συμφορήσεων. Γιατί ενώ θα ταξιδεύουν θα μπορούν να ασχολούνται με άλλα πράγματα οι επιβάτες. Αλλά μπορεί να υπάρξουν και αντικρουόμενα αποτελέσματα γενικά στην κυκλοφορία. Και άρα και στην εκπομπή ε, αερίων καυσαερίου. Γιατί εάν αυξηθεί για αυτούς τους δύο λόγους που ανέφερα στην αρχή η χωρητικότητα του δικτύου μπορεί να υπάρξει περισσότερη κίνηση. Είδαμε και άλλες επιπτώσεις, δεν προλαβαίνω τώρα να σας τις εξηγήσω, αλλά τις ε, βλέπετε σε αυτό είναι εδώ τη διαφάνεια επιπτώσεις στον κλάδο, στην αγορά εργασία, στην ηθική και την δημόσια αποδοχή. Ε, θα έπρεπε παρακαλώ να διαβάσετε τη μελέτη. Ίσως μέσω των ερωταπαντήσεων να πούμε περισσότερα. Ποιες είναι τώρα οι βασικές συστάσεις. Πώς θα αξιοποιήσουμε περισσότερο τις δυνατότητες. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ε, διανομής της γνώσης από τα πιλωτικά προγράμματα και τα τεστ. Επίσης, πρέπει να δούμε την τοπική και αστική άποψη. Γιατί πολλά μπορούμε να επιτύχουμε σε αυτό το επίπεδο, αλλά υπάρχουν και μεγάλοι κίνδυνοι. Υπάρχουν και ενδεχόμενα μειονεκτήματα σημαντικά σε αυτό το επίπεδο. Σε ενωσιακό επίπεδο πρέπει να βρούμε τις διαδικασίες για την οδική κυκλοφορία του μέλλοντος. Πώς θα αλληλεπεδράσουν διάφορα συστήματα. Γενικά υπάρχει νομίζω συνένεση ότι χρειάζεται ένα ενιαίο πλαίσιο πολιτικής ένα ενιαίο πλαίσιο για την αυτοματοποίηση και τη σύνδεση των οχημάτων. Χρειάζεται περαιτέρω διεθνή συνεργασία για τα τεστ για να αξιοποιήσουμε καλύτερα την ε, αυξανόμενη γνώση και για την εισαγωγή στην αγορά σταδιακή προσέγγιση συστήνουμε να ξεκινήσουμε τα χαμηλότερα επίπεδα αυτοματοποίησης που θα μπορούσε να αρχίσουν τώρα να χρησιμοποιούνται και μετά να βασιστούμε σε αυτά για να περάσουμε στα υψηλότερο επίπεδο. Επίσης, στην έκθεσή μα αναφέρουμε μια σειρά οδηγίες που θα έπρεπε να τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν σε αυτή τη διαδικασία για να τη βοηθήσουν. Πολλά από αυτά περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του Άμστερνταμ που γνωρίζετε. Είναι ένα βασικό κείμενο αυτό και ελπίζω οι αναλυτικές μας ε, συστάσεις που είναι στη μελέτη να σας βοηθήσουν στην περαιτέρω εργασία σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Για την παρουσίαση τώρα έχουμε άλλες δύο και μετά ερωτήσεις και απαντήσεις. Στις επόμενες ομιλίες είναι, λιγότερο ο χρόνος, 7 ε, λεπτά το ξέρετε. Και βεβαίως μπορείτε να μιλήσετε και στη μητρική σας γλώσσα, μην διστάζετε. Έχουμε μεταφραστές γι' αυτό. Ε, ο κύριος Στέφαν Νόγκεμπαουερ είναι ε, πρόεδρος της ΕΡΤΡΑΚ της ε, ΜΠΕΜΒΕ. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Με μεγάλη χαρά ήρθαμε να μιλήσουμε για την αυτόνομη αυτόματη οδήγηση. Η κυκλοφορία του μέλλοντος θα είναι διαφορετική από εκείνη που γνωρίζουμε σήμερα. Θα παρακαλούσα να περάσουμε στην παρουσίαση που έχουμε. Βλέπετε εδώ μερικές λέξεις κλειδιά. Ε, η κυκλοφορία του μέλλοντος θα είναι κατά κύριο λόγο ηλεκτρική, διασυνδεδεμένη, διατροπική, αυτοματοποιημένη σε διάφορα μέσα μεταφοράς. Σήμερα συζητούμε την αυτοματοποίηση. Τι περιμένουμε λοιπόν από ε, αυτή την οδήγηση. Τώρα ε, αυτό που βλέπουμε είναι να και προβλέπουμε να αυξηθεί ε, η οδική ασφάλεια. 90% ε, των δυστυχημάτων των τροχαίων προκαλούνται από απροσεξία ή ανθρώπινο σφάλμα. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί. Έχουμε επίσης το πώς θα αποφεύγουμε τα μποτιλιαρίσματα, πώς θα διοχετεύουμε την κυκλοφορία και αντίστοιχη μείωση των καυσαερίων και του διοξιδίου του άνθρακα. Επίσης, ε, όσο ε, γυράσκει και ο πληθυσμός και η κοινωνία μπορούν να οδηγούν και οι μεγαλύτεροι σε άνθρωποι και επίσης ε, αυξάνεται και η δυνατότητα χρήσης του χρόνου του οδηγού και η άνεσή του. Γενικά έχουμε σημαντικές βελτιώσεις. Πότε αναμένεται να γίνει αυτό βέβαια τώρα. Βλέπετε τα διάφορα στάδια της αυτοματοποιημένης οδήγησης δεξιά είναι η πλήρης αυτοματοποίηση, αυτόνομη οδήγηση, το αυτοκίνητο χωρίς οδηγό καθόλου. Και το Google Car δεν θα έρθει ουρανό κατέβατο από τη μια μέρα στην άλλη και θα είναι ταυτόχρονα πλήρως αυτοματοποιημένη η κυκλοφορία στις, ε, στους αυτοκινητοδρόμους. Ε, βλέπετε ε, άλλα συστήματα προειδοποίηση για τις αποστάσεις και ε, διάφορα αυτοματοποιημένα. Βρισκόμαστε δηλαδή μεσούς αυτής της ε, εξέλιξης. Το τι μπορεί να κάνει στο μέλλον ένα αυτοματοποιημένο όχημα είναι ότι κάνει και ο άνθρωπος. Πρώτα θα πρέπει να αντιληφθεί το περιβάλλον, μετά να επεξεργαστεί, να σκεφτεί την πληροφορία αυτή και στη συνέχεια να δράσει. Ε, μέσω από ε, συγκεκριμένα ε, αυτόματα μέσα. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί αισθητήρε για την αντίληψη του περιβάλλοντος. Αυτό δεν είναι μέλλον, αυτό ισχύει. Είναι ένα όχημα που μπορείτε να αγοράσετε και σήμερα, που είναι στην παραγωγή. Στου αισθητήρε ε, που έχει σήμερα ένα σύγχρονο όχημα για υποβοηθούμενη οδήγηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ως εικόνα γιατί μπορείτε να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι για τη δημιουργία αξία και υπεραξία στην Ευρώπη και πόσα μπορεί να κάνει η βιομηχανία και οι προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας, ε, οι αισθητήρε, τα ε, τεχνολογικά Ινστιτούτα, η καινοτομία, όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι πρέπει να μεταφραστούν σε ένα μοντέλο που να μπορεί να λειτουργεί στην πράξη και να έχει νόημα η λειτουργία του. Αυτή λοιπόν η εικόνα, ε, φωτογραφία σας δείχνει τι ευκαιρία έχουμε εδώ για καινοτομία στο μέλλον, για ε, ηγετική θέση της Ευρώπης στην οικονομία και στην απασχόληση. Ε, αυτά τα συστήματα ήδη τα χρησιμοποιούν τα οχήματα και στο μέλλον θα εξακολουθούν να τα χρησιμοποιούν. Και όσο αυξάνεται η ποιότητα της αυτόνομης οδήγησης και της αυτόματης, όσο περάμε σε πιο υψηλά επίπεδα αυτοματοποίησης, τόσο θα χρειαζόμαστε και περισσότερες πληροφορίες από το περιβάλλον γύρω-γύρω. Δηλαδή, εδώ μιλάμε συστήματα τηλεπικοινωνίας ε, και πληροφορίες που θα έρχονται επιπλέον στο αυτοκίνητο. Και αυτό είναι το δεύτερο σημαντικό που θέλω να τονίσω. Άρα, χρειαζόμαστε κάλυψη ε, τηλεπικοινωνίας ε, σε όλη την επικράτεια, σε, σε όλη τη διαδρομή. Και κυρίως επειδή η αυτόματη οδήγηση έχει πολύ μεγάλη σημασία ε, να γίνεται σε μεγάλες επεφάνειες, δηλαδή ε, στην Ήπεθρο, σε αυτοκινητοδρόμους. Χρειαζόμαστε λοιπόν την τεχνολογία ε, στην Ήπεθρο, σε όλη την επικράτεια και, και συνήθως τηλεπικοινωνίες οι οργανισμοί ενδιαφέρονται για τα αστικά κέντρα και όχι για την Ήπεθρο. Για τις συγκοινωνίες και για τις μεταφορές όμως θα πρέπει αυτό να γίνει στην Ήπεθρο. Στη συνέχεια, είναι πολλά τα στοιχεία αυτά ε, που θα πρέπει να επεξεργάζεται το όχημα σε πραγματικό χρόνο. Και η τηλεπικοινωνία και η επικοινωνία στο όχημα θα πρέπει να είναι ασφαλής. Αυτό είναι πρόκληση κυρίες και κύριοι, για να το πω ξεκάθαρα. Υπάρχουν ορισμένοι που ισχυρίζονται ότι το αυτοκίνητο του μέλλοντος ε, είναι ένα κινητό με τέσσερις τροχούς. Ε, δεν είναι έτσι όμως. Ένα κινητό τηλέφωνο. Ε, είναι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να είναι ένα τηλέφωνο, smartphone ε, με τέσσερις ε, τροχούς. Τελείως διαφορετική είναι η αίσθηση και αντίληψη ασφάλειας. Ποτέ των ποτών δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Ε, πόσο καιρό χρησιμοποιείτε το κινητό σας, αυτό που έχετε τώρα, δύο χρόνια, τρία χρόνια, πέντε, δέκα. Γιατί ρωτάω για τη δεκαετία. Γιατί είναι ο μέσος όρος ε, ενός, ηλικίας ενός οχήματος στην Ευρώπη. Δηλαδή ο κόσμος έχει αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην αγορά έχει 10 και 20 χρόνια και θα πρέπει να εγγυηθούμε την ασφάλεια για 20 και πλέον έτη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η διαφορά με την ε, βιομηχανία κινητών τηλεφώνων, ε, smartphone. Εμείς λοιπόν ως κλάδος θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα όχημα που να έχει ασφαλής τηλεπικοινωνίας. Ακριβώς δεν θα πρέπει οποιοδήποτε να συνομιλεί ας πούμε με το αυτοκίνητο. Θα πρέπει να γίνουν δομές, ε, πλατφόρμες ασφαλείς η πλατφόρμα μπορεί να μιλάει και με το Θεό τον ίδιο, αλλά το αυτοκίνητο ε, θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο συνομιλήτη. Yeah. Επίσης χρειαζόμαστε προνομιούχες επικοινωνίες, τηλεπικοινωνίες ε, μέσα στο όχημα, γιατί αν υπάρχει και σύστημα προειδοποίησης για κινδύνους, ε, αυτά τα, τα σήματα θα πρέπει να εκπέμπονται σε πραγματικό χρόνο και άμεσα. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται σε ένα περιβάλλον που εμφανίζονται νέοι ε, φορείς και παίκτες εντό εισαγωγικών στο διεθνές στερέωμα. Για να μιλήσω μόνο για την αυτόνομη ή αυτόματη οδήγηση, κοιτάξτε πόσοι ενέχονται εδώ. Βεβαίως η αυτοκινητομηχανία, οι κατασκευαστές, οι προμηθευτές τους, αλλά και η κοινωνία που να είναι πρόθυμη να το υιοθετήσει αυτό. Χρειαζόμαστε νομοθέτες, κοινοβούλια και ο καθένας έχει το ρόλο του, που είναι και σημαντικός. Και φυσικά χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες για την ανταλλαγή των δεδομένων. Εδώ μπαίνουν λοιπόν οι νέοι ε, παίκτες, όπως είναι οι αμερικανικές εταιρείες, Google, Apple κλπ, που έχουν μεγάλη πείρα στη διαχείριση μεγάλων και πολλών δεδομένων και έχουν και μεγάλη οικονομική ισχύ. Για να καταλάβετε την τάξη μεγέθους, έχουν πολύ ε, περισσότερα χρήματα αυτές οι αμερικανικές εταιρείες από ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Συνοψίζω, ε, η τεχνολογία αυτή είναι μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη, ε, για την απασχόληση, για την κοινωνία, για το περιβάλλον, για την κυκλοφορία. Είναι τεράστιες οι προκλήσεις και στη βιομηχανία λοιπόν και στην κοινωνία. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει ε, ένα πάρα πολύ σωστό πρόγραμμα έρευνας και νοτομίας για να παραμείνουμε ηγετική δύναμη παγκοσμίω. Εμείς ως πλατφόρμα τεχνολογίας ασχολούμαστε εντατικά και έχουμε και τον πρώτο το οδικό χάρτη ε, που ενημερώνεται ε, κάθε φορά που έχουμε νέες εξέλιξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Νόγκεμπάουα. Και τώρα ο κύριος Μπέτ Μίλλερ από την εταιρεία Carpostal, την ελβετική εταιρεία δημοσίου μεταφορών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με τα χαράς να σας παρουσιάσω και τη δική μας την άποψη και την ε, σύντομη εμπειρία μας για κάτι που μόλις ξεκινήσαμε. Δύο λόγια για την επιχείρησή μας που μπορεί να μην είναι γνωστή σε όλους. Έχουμε πάνω από 100 χρόνια εμπειρίας ε, στις δημόσιες μεταφορές. Ε, αρχίσαμε να μεταφέρουμε κόσμο στα ελβετικά ε, και το κάνουμε ακόμα και σήμερα. Ε, στην Ελβετία, στο σύνολό της και επίσης και στη Γαλλία και στο Λίχτενστάιν και προσφέρουμε ε, συνδυασμένες μεταφορές. Ε. Υπάρχουν λοιπόν και άλλες υπηρεσίες, συμπληρωματικές στις υπηρεσίες που προσφέρουμε στην Ελβετία. Το θέμα μας βέβαια είναι η εμπειρία που είχαμε με τα ε, αυτόνομα αυτά οχήματα. έχουμε ένα όχημα εννέα θέσεων, είναι μικρή εικόνα, δύο μάλιστα τέτοια οχήματα που είναι σε μια μικρή πόλη στη Σίων, γι' αυτό και τη λέμε και την εμπειρία του Σίων. Πρόκειται για ευφυή οχήματα, τα οποία είναι πλήρως αυτόνομα. Και θα χρησιμοποιηθούν στους δρόμους της πόλης από τον Ιούνιο φέτος. Και θα μεταφέρουν κόσμο φυσικά σε αυτή τη μικρή πόλη στην Ελβετία. η ιδέα είναι να χρησιμοποιούν αυτό το μικρό ε, λεωφοριάκι όλοι, οποιοδήποτε βρίσκεται στη στάση του λεωφορείου. Θα υπάρχει όμως και μία εφαρμογή ε, on demand που θα μπορεί κάποιος να καλέσει αυτό το όχημα κατόπιν ετήματος. δεν θα είναι ε, εντελώ ανοιχτή περιοχή, θα περιορίζεται στους δρόμους της πόλης της Σιών και θα περιλαμβάνει κάθε δρόμο, ε, συνηθισμένους δρόμους που υπάρχει συνηθισμένη κίνηση, ε, εσωτερικούς ε, δρόμους με ε, πλακάκια και στο μεγάλο, στην ανηφόρα, στο τουριστικό σημείο της πόλης θα μπορεί μάλιστα να κάνει και κάποια παράκαμψη το όχημα και να ακολουθήσει μια διαφορετική διαδρομή από αυτήν που είναι στην προκαθορισμένη περιοχή που θα κυκλοφορεί. Δεν θα το κάνουμε αυτό μόνοι μας βέβαια. Συνεργαζόμαστε με πανεπιστήμια, με το Πανεπιστήμιο της Λοζάνης ε, κυρίως, το UPFL και άλλα ακαδημαϊκά Ινστιτούτα και χρησιμοποιούμε ένα όχημα το οποίο κατασκευάζεται από μια γαλλική νεοφυή επιχείρηση έχει ένα λογισμικό ελέγχου, το οποίο κατασκευάζεται από μια άλλη μικρή επιχείρηση στην Λοζάνη. Πρόκειται λοιπόν για ένα αμυγός ευρωπαϊκό ε, πρόγραμμα. Είναι ένα όχημα λοφοριάκι, το οποίο έχει κατασκευαστεί από ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και πιστεύουμε ότι αυτά τα αυτόνομα οχήματα, ιδίως αυτά τα μικρά λοφοριάκια, θα μπορούν να ε, έρθουν να προσθεθούν στις δημόσιες συγκοινωνίες μας, ε, να είναι το τελευταίο ή το πρώτο κομμάτι μιας διαδρομής από τις βασικές ε, γραμμές λεωφορείων και τρένων που έχουμε. Κάτι άλλο το οποίο θα δοκιμάσουμε εδώ στο Ισιόν είναι οι μεταφορές τουριστών. Οι οποίες φυσικά ποικίλουν ανάλογα με την εποχή και το καιρό να υπάρχουν φυσικά και άλλες χρήσεις, να τα χρησιμοποιεί κάποιος ε, για να πάει για ψώνια ή κάποιες σύντομες διαδρομές για να μπορέσουν ε, να κουβαλήσουν τα ψώνια τους. Αυτές είναι οι βασικές εφαρμογές ε, που θεωρούμε ότι θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα οχήματα για την επόμενη διετία και από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα μπορέσουμε να έχουμε κάποιες περαιτέρω εφαρμογές που θα ενισχύσουν τις δημόσιες μεταφορές μας η άποψή μας, το όραμά μας ε, από το τομέα των δημοσίων μεταφορών και εδώ μιλώ και εξ ονόματος ε, του συνδικάτου μας, του UATP, ε, γιατί είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Μεταφορών, πιστεύουμε ότι αυτά τα οχήματα μπορούν να έρθουν να προσθεθούν στις υπηρεσίες που παρέχουμε για τις δημόσιες μεταφορές και το όραμά μας, όπως σας είπα, δεν είναι ε, να έχουμε αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς στους δρόμους, να έχουμε οδηγούς χωρίς αυτοκίνητο. Διότι το βασικό πρόβλημα με τα αυτοκίνητα τα ιδιωτικής χρήσεως είναι ότι ε, οδηγούν σε κυκλοφοριακή συμφόρηση και αυτό είναι φυσικά ένα πρόβλημα το οποίο θα αυξηθεί με την αύξηση του πληθυσμού. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μπορούν ακόμα να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο οι δημόσιες μεταφορές και μπορούν να βελτιωθούν έτσι περαιτέρω και να είναι πολύ πιο αποτελεσματικές ε, και επομένως να τις χρησιμοποιούν περισσότεροι, χρησιμοποιώντας κυρίως αυτή την τεχνολογία στην οποία ε, δοκιμάζουμε για αυτά τα νέα προϊόντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για αυτές τις τρεις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Και τώρα ο Βιμ Φαντακάμπ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. I will speak in Dutch. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Um, Πρώτον, Πρόεδρε, έχω μια διοικητική ερώτηση. Έχουμε τρεις εκθέσεις λάβει, αλλά όχι την έκθεση κυρίας Φριζόνη. Θα μας τη δώσετε ή μας φτάνουν αυτά. Καμία σχέση βέβαια οι τρεις εκθέσεις με αυτά που είπε η κυρία Φριζόνη. Τη δική της έκθεση τι θα την κάνετε. Ερώτηση δεύτερη προς τον κύριο Νόιγκεμπάουα. Και έχει να κάνει με το εξής. Τα πέντε επίπεδα. Είπατε ότι είμαστε κάπου στη μέση τώρα. Ο κύριος Κράμερ και εγώ την περασμένη εβδομάδα πήγαμε στο Συμβούλιο στο Άμστερνταμ που μας είπαν ότι είμαστε στο τέλος περίπου της δεύτερης φάσης. Εσείς λέτε ότι είμαστε στη μέση. Γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και επίσης, ρωτώ, θα φτάσουμε ποτέ στο επίπεδο 5 και αν ναι, πότε προβλέπετε περίπου. Και ρωτήσω και τον κύριο Μιούλαφ, αν το λέω καλά. Την χάνει να γνωρίζω την πόλη της Σιών. Έχω πάει διακοπές και στο Μπρίκ και στο βίσκο και στη Σιόν είναι πολύ ήσυχο Έχει ωραίες εκκλησίες και όλα τα συμπαραμαρτούντα. Εκεί υπάρχει αρκετή διάδραση με ξέρω παιδιά, πεζούς που περνάνε απέναντι, του διασχίζουν δρόμους, τουρίστες για να δοκιμάσετε ε, αυτό το λεωφοριάκι. Γιατί δεν το κάνετε στο κέντρο της Γενέβης ή της Βέρνης για παράδειγμα. Ευχαριστώ ο Ισμαήλ Ερτούκ. Δυστυχώ πρέπει να σας διακόψω τη συνομιλία σας. Ευχαριστώ για τη μελέτη και για τις παρουσιάσεις. Η αυτοματοποίηση είναι ένα από τα χόμπι μου και θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει τα τελευταία χρόνια και δεκαετίες για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την εισαγωγή του ως πολιτική. Δεν θα πω τίποτα για αυτά που αναμένω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι, ότι στον ορίζοντα 2020, το πρόγραμμα ορίζοντα 2020, προβλέπονται 20 εκατομμύρια 100 συγγνώμη εκατομμύρια για τις οδικές μεταφορές. Καλό αυτό. Αλλά να μην βιαστούμε να χαρούμε πάρα πολύ. Γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε διαθέτουν τέσσερα δις. Είναι θέματα τάξης μεγέθους. Αλλά εν πάση περιπτώσει καλό είναι να έχουμε κάποιες χρηματοδοτήσεις. Ξέρω ότι η ευρωπαϊκή πολιτική υστερεί. Δεν είμαστε στο επίπεδο που θα έπρεπε να είμαστε. Και μα, θα πρέπει να το δούμε σοβαρά. Μήπως θα έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα ειδικό χρηματοδοτικό μέσο για την ψηφιοποίηση των μεταφορών. Γι' αυτό, αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσουμε ένα σαφές νομικό πλαίσιο που να λύσει όλα αυτά τα ανοιχτά θέματα που ήδη αναφέρθηκαν και άλλα που θα αναφερθούν, προστασία των δεδομένων, κυβερνοασφάλεια, ασφάλεια των οδηγών μεταφορών και επίσης να υπάρξουν και επαρκείς χρηματοδοτήσεις. Θα ήθελα να κάνω κάποιες τεχνικές ερωτήσεις. Γιατί το πρώτο θέμα που πάντα τίθεται είναι ότι αν δεν χρειάζεται να βάλουμε τα χέρια στο τιμόνι και στο μοχλό και τα λοιπά Τι θα γίνει αν παρόλα αυτά προκύψει ένα ατύχημα. Όχι από πλευράς ευθύνη, αλλά τεχνικά δηλαδή. Όχι από πλευράς ε, ασφάλισης αλλά τεχνικά διότι ξέρουμε ότι τα διάφορα συστήματα ραντάρ, βοήθησης και οι κάμερες μπορούν να παρέμβουν. Και πόσο αξιόπιστα είναι. Και αν υπάρξει μια κατάσταση ανάγκης, ο οδηγός μπορεί να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη. Υπάρχει συζήτηση με, με τιμόνι χωρίς τιμόνι. Ορισμένοι λένε δεν χρειάζεται τιμόνι. Άλλοι λένε όχι, όχι, πρέπει να υπάρχει τιμόνι γιατί μπορεί να χρειαστεί να παρέμβει ο οδηγός να πάρει το τιμόνι. Πρέπει να υπάρχει για να το πάρει. Ε, πολύ ενδιαφέρον αυτό, με ενδιαφέρει. Και κάτι άλλο. Πόσο πιθανό είναι να υπάρξει ένα λάθος προγραμματισμού το οποίο να σημαίνει ότι εκατομμύρια οχήματα που να έχουν ένα πρόβλημα και δεν είναι ε, εύκολο να τα, να, να, να τα όλα αυτά. Άρα είναι τεράστιος ο κίνδυνος. Ευχαριστώ. Ντομινίκ Ρικέου επόμενος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εθίγησα μια σειρά αποζητήματα. Διαπιστώνουμε ότι έχει υπάρξει πρόοδος και ότι έχουμε δυνατότητα να περάσουμε από τη δεύτερη και τρίτη προς τις παραπάνω κατηγορίες. Αλλά μία ερώτηση που θέλω να, δέσω στους, να θέσω στους τρεις παρεμβαίνοντες εκπλήσωμε από το πόσο χρόνο θεωρούν ότι χρειάζεται για να φτάσουμε στην κατηγορία 5. Ακόμη 20 χρόνια για να φτάσουμε στην κατηγορία 5. Αλλά αν δω πόσο χρόνο χρειαστήκαμε για να φτάσουμε από το 0 στο σημερινό επίπεδο, λίγα χρόνια, ούτε καν δεκαετία. Γιατί λοιπόν θέλουμε τόσο χρόνο, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ε, τα νέα μοντέλα τέτοιων οχημάτων ή θεωρείτε ότι θα είναι κυρίως η υποδομή που θα χρειαστεί να αναπτύξουμε και ότι θα χρειαστούν γι' αυτό και, περίπλο, και περίπλοκες τεχνολογικές εξελίξεις για να υπάρχουν οι αναγκαίες επικαλύψεις ή θεωρείτε ότι θα πρέπει να κάνουμε μεγάλες επενδύσεις επί των ε, υποδομών. Και δεύτερη ερώτηση. Η ανάπτυξη αυτών των ε, αυτοοδηγούμενων οχημάτων θα πρέπει καταρχάς να εισαχθεί στις πόλεις όπως γίνεται τώρα σε συγκεκριμένα δρομολόγια ε, που είναι κλειστά για κάθε άλλου είδους κυκλοφορία όπως στη Σιόν και στη Λαγοσέλ ή θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στους μεγάλους οδικούς άξονες. Δηλαδή, εκεί που υπάρχει περίπλοκη μεικτή κυκλοφορία, δηλαδή άλλα οχήματα, πεζή κτλ. Εκεί πρέπει πρώτα να επιδιώξουμε να εισαγάγουμε αυτό το πράγμα ή θα πρέπει κυρίως να στραφούμε προς τις ε, δημόσιες μεταφορές και συγκοινωνίες μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων. Θέτω λοιπόν το ερώτημα. Πόλεις, μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις ή το όχημα που θα αναπτυχθεί θα μπορεί να τα κάνει όλα. Θα μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικό και σε αστικές περιοχές και σε ε, υπεραστικές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η Καρίμα Ντελή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είμαι και συγκίτρια για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, αλλά όχι μόνο αυτό, γιατί τι κάνουμε τώρα για τον 21ο αιώνα, ε, εφευρίσκουμε ε, τα δικαιώματα των ρομπότ. Πόσο θα κοστίσει δηλαδή ένα αυτόνομο όχημα, πόσο κοστίζει σήμερα ή πόσο θα μας κοστίσει. Δεύτερη ερώτηση. Συμφωνώ με τον Ντομινίκ και Έχουμε εξάρτητα οχήματα, διασυνδεδεμένα ήδη, που θα έρχονται σε 10-15 χρόνια. Τώρα θα έχουμε και το αυτόνομο όχημα. Και ποιος φέρει την ευθύνη σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματο. Αφού δεν θα υπάρχει οδηγό, τι θα πταίει, ο κατασκευαστή, η ε, υπάροχη του διαδικτύου, ποιο, δεν ξέρω. Ε, Ω νομοθέτες εμεί τώρα τι καλούμεθα να αποφασίσουμε, Ποιο θα έχει την ευθύνη. Έχετε προτάσεις για την ευθύνη. Είδαμε το σκάνδαλο της Volkswagen στη συνέχεια. Και τι μας είπανε ότι πολλοί κατασκευαστές δεν τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Και συχνά και έμεσα ποιος την πληρώνει, ο πολίτης. Αυτό το ζήτημα της Volkswagen φωτίζει και το θέμα αυτό του αυριανού αυτοκινήτου. Και ποιος θα δώσει την έγκριση για τους τύπους αυτοκινήτων αυτών. Πώς θα γίνει. Ποιος θα δώσει την άδεια για να κυκλοφορούν στην αγορά και στους δρόμους μας αυτά τα νέα αυτοκίνητα. Α, χρειαζόμαστε ε, νέο ευρωπαϊκό οργανισμό. Άλλον ένα για το αυτοκίνητο του αύριο. Αυτό σας ερωτώ. Βεβαίω, λογικά, μιλήσατε πάρα πολύ για το κλίμα και ως εισηγήτρια για τη βιώσιμη αστική ε, κινητικότητα, μπορώ να σας πω ότι το διασυνδεδεμένο αυτοκίνητο δεν πρόκειται να υποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει τα αυτοκίνητα που ήδη κυκλοφορούν. Θα προσθεθεί άλλο ένα είδος οχήματος. Και προσοχή, να μην παραγωνιστούν τα αυτοκίνητα. Ακόμα και αν δώσατε αυτή την ε, η πρόταση, κάνατε αυτή την επίδειξη για το λεωφορείο του αύριο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα μαζικά μέσα επικοινωνίας. Και επίσης τι θα καίνε από καύσιμο. Θα είναι όλα ηλεκτρικά αυτά τα αυτοκίνητα. Ε, δίζελ. Πετρέλαιο. Ή έχετε αποφασίσει να ε, εφεύρετε και τα νέα καύσιμα του μέλλοντος. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, ε, πρόεδρε τρο, Τροχάδη, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι. Αλλά το ουσιαστικό ερώτημα, έχω άλλα δύο, τι γίνεται με την προστασία των δεδομένων. Ακροθυγός την αναφέρατε. Αυτό είναι τεράστια υπόθεση. Και ένα τελευταίο. Θα είπε και ο συνάδελφος μου, Ντομινίκ Χρικέ. Για να έρθει το συνδεδεμένο αυτοκίνητο θα πρέπει να ερωτήσετε τη ΣΟΤΑ, τις, ε, τους Δήμους ε, χρειάζεται και ένας νέος κόκ, ε, κώδικας ειδικής, οδικής συγγνώμη, <laughs> κυκλοφορίας, κυκλοφοριακά σχέδια. Πώς θα τα αριθμίσετε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ο Πέτερ Λούντγκρεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η ιδέα ενός αυτοκινούμενου οχήματος που χωρίς οδηγό ε, πραγματικά με τρελαίνει. Ε, όπως όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να οδηγώ και πραγματικά μισώ την ιδέα να αποφασίζει το αυτοκίνητο για μένα και να μην μπορώ εγώ να ελέγξω το αυτοκίνητο. Παραδείγματο χάρη, κάθεστε σπίτι σα στον υπολογιστή σα μπροστά και τι γίνεται άμα χαλάσει ο υπολογιστή, δεν λειτουργεί τίποτα, πρέπει να τον κλείσετε, να ξανακάνετε reboot από την αρχή. Εγώ δεν θέλω να βρεθώ σε αυτοκίνητο και να του συμβεί κάτι τέτοιο, αν ξαφνικά εντό εισαγωγικών ε, ε, κρασάρει το σύστημα. Τώρα, για να είναι βιώσιμο από οικονομική σκοπιά ε, ένα τέτοιο ε, πρόγραμμα, πρέπει ε, να ε, πείσουμε τους ανθρώπους και αν ε, τους πιέσουμε δεν θα είναι επιτυχία. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα τα αγοράσει. Πρέπει να είναι ελεύθερη επιλογή να χρησιμοποιήσει κάποιος αυτή τη μέθοδο. Σε αυτούς που αρέσει να οδηγούν το αυτοκίνητο θα πρέπει να δίνεται το ελεύθερο να οδηγούν τα αυτοκίνητά τους στο μέλλον και αν ε, δεν νιώθει κάποιος ασφαλής σε ένα αυτοκίνητο το οποίο το οδηγεί ένα σύστημα καλωδίων τότε να αφήνει το αυτοκίνητο να οδηγεί γι' αυτόν. Δεύτερον, ασφάλεια. Ποιο θα πληρώνει την ασφάλεια, ποιο θα καλύπτει το κόστο ε, εάν συμβεί κάτι. Και επίση θα ήθελα να ξέρω εάν υποχρεώσετε τον κόσμο να χρησιμοποιεί μια τέτοια λύση, ε, τι θα κάνετε, θα του υποχρεώσετε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόχ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Προς την ίδια κατεύθυνση και η δική μου ερώτηση. Εμένα η τεχνολογία πραγματικά με συναρπάζει και τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης που έχουμε σήμερα με ενθουσιάζουν, αλλά το συζητάω με πολίτες και βλέπω ε, ήδη αντίσταση και μεγάλη αγωνία ε, ότι θα γίνει αν ε, κρασάρει και αν χακάρει κανείς το σύστημα. Στην ΠΕΜΒΕ, ξέρετε, το έχετε και ως επιχείρημα διαφήμιση για τα αυτοκίνητα ότι αρέσει στον οδηγό να οδηγεί ένα BMW. Ευχαριστώ να σας πω καταρχάς ότι εγώ δεν φοβάμαι αυτό την οδήγηση χωρίς αυτοκίνητο. Ε, ίσως θα ήθελα να σας πω να μας βάλετε να τη δοκιμάσουμε γιατί ο καθένας θα ξεπεράσει και τους φόβους του έτσι. Επίσης να σας πω ότι στην πλειοψηφία των ε, αεροπορικών πτήσεων το μεγαλύτερο τμήμα γίνεται αυτομάτως και κανένας δεν τρομάζει για κάτι τέτοιο. Ε, έχω κάποιες πρακτικές αμφιβολίες. Η αυτόματη οδήγηση προϋποθέτει κάποιες υποδομές που σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν και δημόσιες επενδύσεις. Ε, όχι μόνο ε, κάποιου αισθητήρε ε, και κάποια καλώδια, να υπάρχει κατάλληλη δυνατότητα διασύνδεσης. Εμείς στην πλειοψηφία της Ευρωπαϊκής Επικρότειας δεν έχουμε καν ευρυζωνικές υπηρεσίες. Επομένως, ε, δεν θα πρέπει να ρωτάμε σε πόσο χρόνο μπορούμε να έχουμε τα αυτοκίνητα, αλλά σε πόσο χρόνο μπορούμε να έχουμε τις κατάλληλες υποδομές για να υποστηρίξουν τα αυτοκίνητα. Επίση, δεύτερον, έχουμε το θέμα τη ευθύνη. Όντω εδώ έχουμε μια φαιά ζώνη. Ε, έχουμε βασιστεί αυτή τη στιγμή στην ε, ε, έννοια της υποκειμενικότητας, της προσοχής του οδηγού. Προσαρμόζεται στις κλιματικές συνθήκες, τα εμπόδια που αντιμετωπίζει, τις δυνατότητες που έχει και το αυτοκίνητό του. Επομένως υπάρχει μια προσωπική επιρροή και από εκεί και πέρα ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη και αυτό το καλύπτει το νομικό πλαίσιο. Αύριο, εάν συμβεί κάτι, ε, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, ο συντηρητής, ε, η σύνδεση του δικτύου, το εμπόδιο το οποίο μπορεί να προκύψει ξαφνικά, ποιος θα είναι ο υπεύθυνο. Νομίζω ότι αυτό θα τρομάξει τον καταναλωτή όταν θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσο θα πρέπει να αγοράσει ένα τέτοιο όχημα. Σίγουρα υπάρχουν εξαιρετικές ευκαιρίες. Ε, πολλοί άνθρωποι θα μπορούν να είναι πλέον πιο αυτόνομοι χρησιμοποιώντας τέτοια αυτοκίνητα αλλά αναρωτιέμαι τι γίνεται με το κόστος. Ε, μας χρειάστηκαν 20 χρόνια για να έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία μπορεί κάποιος να αγοράσει. Ίσως το μέλλον δεν θα είναι απλώς η αγορά, αλλά ίσως ε, στη βιομηχανία 4.0 να είναι η αγορά της υπηρεσίας αυτή η οποία θα λαμβάνεται υπόψη. Αναρωτιέμαι λοιπόν κατά πόσο νομίζετε ότι αυτό θα είναι το μέλλον που μας περιμένει και εάν θα έχουμε οχήματα όχι σαν τα παραδοσιακά που γνωρίζουμε σήμερα, αλλά σαν αυτά που έδειχναν πριν από κάποια χρόνια κάποια ε, περιοδικά, κάποια φουτουριστικά αυτοκίνητα, μονοθέσει αυτοκίνητα, τα οποία θα μπορούσαν ίσως να προσαρμοστούν ε, και να έχουν και άλλες θέσεις για τους που σαν ε, χρειαστεί. Κύριε... Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο θέματα. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, ο κύριος Νόγεμπάουερ αναφέρθηκε στην έννοια του διασυνδεδεμένου αυτοκινήτου. Αυτό που με ενδιαφέρει ένα πρωτίστως σκεπτόμενος και τα συστήματα τα οποία που χρησιμοποιούν οι διάφοροι κατασκευαστέ είναι ε, κατά πόσον είναι συμβατά αυτά τα συστήματα μεταξύ τους. Αναφερθήκαμε σε έξυπνα τηλέφωνα, σε υπολογιστές. Υπάρχει ε, κάτι αντίστοιχο με τη συζήτηση Windows, Android, ε, Apple, δηλαδή υπάρχουν αντίστοιχα συστήματα που μπορεί να μην είναι συμβατά μεταξύ τους. Και επίσης, τι θα γίνει ε, στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας από πλευράς καινοτομία, ώστε να μην συμβεί αυτό το οποίο συνέβη στην Νόκια. Ξέρουμε όλοι τι έγινε. Η Νόκια έζησε τη χρυσή εποχή της κινητής τηλεφωνίας κάποια στιγμή και μετά ε, είχαμε εξελίξεις από άλλες περιοχές και επιβλήθηκαν τα δικά τους τα τηλέφωνα. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να συμβιβάσουμε την πτυχή της ε, καινοτομίας και στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Άλλη ερώτηση. Σε περίπτωση ατυχήματος, από πλευράς ασφάλειας τι συνέπειες θα υπάρχουν, τι είδους ασφάλιση πρέπει να διαθέτει κάποιος. Εγώ ακόμα δεν έχω μιλήσει με ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά πώς προετοιμάζονται οι ασφαλιστικές εταιρείες για αυτό το μεγάλο μήνα. Μαρίντελβο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ακρόαση αυτή. Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής σας. Είμαι μέλος της Νομικής Επιτροπής και προεδρεύω μιας ομάδας εργασίας για τις νομικές και ηθικές επιπτώσεις της ρομποτικής. Και από αυτή την ε, άποψη ενδιαφέρομαι για τις ε, επιπτώσεις ε, σε αυτά τα θέματα των οχημάτων χωρίς οδηγό γιατί τα, που μπορούν να θεωρηθούν ρομπότ. Και συζητάμε λοιπόν για θέματα ευθύνης, ασφάλισης και μια έκθεση πρωτοβουλίας θα υποβληθεί τέλη Μαΐου και ελπίζω η Επιτροπή σας να συμβάλλει όταν θα διανεμηθεί το σχέδιο έκθεσης. Πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Συμφωνώ βέβαια με όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Μία πολύ συγκεκριμένη ερώτηση για τον κύριο Μούλα. Η προσπάθεια αυτή στην Σιόν. Καταλαβαίνω πως είναι πολύ απαιτητική για την τεχνολογία, την επικοινωνία, την ανταλλαγή δεδομένων. Η πόλη της Σιόν χρειάστηκε να εγκαταστήσει ειδικέ υποδομές για να μπορούν να κυκλοφορούν αυτά τα λεωφορεία χωρίς οδηγό. Γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν παντού αυτά τα λεωφορεία. Γιατί? Για λόγους έτσι δρομολογίου ή γιατί δεν υπάρχουν παντού οι δομές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, και ευχαριστώ για την παρουσία των ομιλητών αλλά ευχαριστώ και για τη δική σας παρουσία γιατί αποδεικνύει ότι αυτά που κάνουμε ενδιαφέρουν και άλλες επιτροπές και χαίρομαι που ήρθατε στην επιτροπή μας και σίγουρα θα συνεχίσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας. Ζωγς Μπαχ Ευχαριστώ. Οι Λουξεμβουργέζοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται για όλα. Δεν είμαστε βέβαια ιδιαίτερα πολλοί, αλλά είμαστε αποτελεσματικοί. Πολλοί συναδελφοί έθεσαν ήδη ερωτήματα για την ε, αστική ευθύνη και καταλαβαίνω ότι θα είναι περίπλοκο. Ξέρουμε ότι αν υπάρξει κάποιο τεχνικό πρόβλημα ανακαλούνται τα οχήματα και τι δύσκολο να καταλάβουμε τι κρύβεται από πίσω και, πώς να, και πόσο προσπαθεί ο κλάδος να μην παραδεχθεί την ευθύνη του κτλ. Άρα πείτε μας για αυτό το θέμα ευθύνης, αστικής ευθύνης. Δεύτερον, η ευελιξία. Το αυτοκίνητο αλλά και τα φορτηγά για μένα έχουν το τρομερό πλεονέκτημα ότι είναι ευέλικτα έναντι των οχημάτων που πρέπει να κινούνται κατά μήκο ε, γραμμών, δηλαδή τα τρένα και τα τραμ. Θεωρώ ότι για τεχνικούς λόγους που έχουν να κάνουν και με το αυτοκίνητο αλλά και με την υποδομή, θα χαθεί ένα μεγάλο τμήμα αυτή τη ευελιξία, τη δυνατότητα να μετακινηθούν παντού. Ισχύει αυτό. Είναι σκόπιμο. Πώ αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα, αυτό το περιορισμό αυτή τη μεγάλη ε, κινητικότητα των οχημάτων. Κάτι που έχει να κάνει και με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι Κόχ και Ντέλη. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν ανησυχίες και φόβοι των οδηγών έναντι του ενδεχομένου βλάβης ή του ενδεχομένου hacking. Και αυτό που είπε και η κυρία Ντέλη, αυτή η ευρωπαϊκή συνεργασία. Βλέπουμε ότι οι κυριότερες αυτοκινητοβιομηχανίες ε, κάνουν η κάθε μία το δικό της και ε, η κάθε μία ε, ε, αναπτύσσει νέα προϊόντα. Δεν υπάρχει επαρκή συνεργασία. Θα ήταν δυνατόν να υπάρξει συνεργασία όπως είχαμε στην περίπτωση του Airbus. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Τώρα να μιλήσω κι εγώ. να μπορέσουν να απαντήσουν οι ομιλητές μας τα αυτοματοποιημένα αυτοκίνητα δεν είναι τίποτα καινούριο. Εγώ ε, κατάγομαι από το Βερολίνο, το έχω ξαναπεί. Πριν από 30 χρόνια είχαμε αυτοματοποιημένο μετρό. Ήταν η γραμμή 4. Ε, δεν είχε οδηγό, αλλά δεν έμπανε και ψυχή μέσα. Βάζανε λοιπόν ένα οδηγό που δεν έκανε τίποτα, απλώς τον έβλεπαν οι επιβάτες, ότι εκεί κάθεται ένας που δεν οδηγούσε. Τα πάντα ήταν αυτόματα και στη Λίλη το μετρό αυτόματο είναι, τίποτα δεν είναι καινούριο. Το καινούριο είναι αυτοματοποιημένα οχήματα. Και ε, το καλύτερο που άκουσα σήμερα ήταν ε, αυτό που θέλουμε ε, είναι από τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό να περάσουμε σε οδηγούς χωρίς αυτοκίνητα. Είπατε ότι μέσο όρο ζωής ε, είναι μια δεκαετία, καλά παραπάνω, εντάξει, κατά μέσο όρο, αλλά ε, ε, κάθε αυτοκίνητο κινείται μία ώρα την ημέρα. Τις υπόλοιπες 23 είναι παρκαρισμένο. Εάν το καταφέρουμε αυτό να έχουμε οδηγούς χωρίς αυτοκίνητα θα μειωθεί ο στόλος. Αυτό είναι επικίνδυνο βέβαια για την αυτοκινητοβιομηχανία. Θυμάμαι ε, στο Μόναχο μία ε, περίπτωση που ήταν συνέδριο και ε, και είχε πει ο δήμαρχος τότε του Μονάχου ότι BMW στο μέλλον σημαίνει στα αγγλικά το είπε ποδήλατο, μετρό και βάδισμα. Ε, και το βρήκα πολύ θέρα, λέω, για ε, το Μόναχο που είναι η έδρα της BMW. Ε, πώς μπορείτε να σώσετε τις θέσεις εργασίας, θα το δείτε βέβαια. Και πριν από 25 χρόνια η Daimler-Benz δεν έφτιαχνε μόνο Mercedes, ε, αλλά και προαστηγακό σιδηρόδρομο, Intercity, μέχρι και ποδήλατα και λεωφορεία και φορτηγά. εάν επιβληθούν ε, τα αυτόματα οχήματα ε, θα επικρατήσουν και στις δημόσιες συγκοινωνίες και ε, κλασικό παράδειγμα αυτό που ακούσαμε από την Ελβετία. Θα υπήρχε η ανάγκη να αλλάξει νοοτροπία και τακτική και η αυτοκινητοβιομηχανία και να προχωρήσει για να συμμετέχει στο μερίδιο και άλλων μέσων μεταφοράς που θα είναι πλέον αυτόματα για να σωθούν θέσεις εργασίας. Αυτό είναι αχαλήνοτη και ανόητη φαντασία δική μου ή έχει νόημα. Ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Πρώτη κυρία Φρυσόνη. Thank you. Yeah. Ευχαριστώ. Ναι. Many different uh, ideas. Uh, Πολλές και διάφορες ιδέες και προτάσεις ακούσαμε θα προσπαθήσω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις και μετά να αφήσω το λόγο για τους υπολείπους, γιατί πολλές από τις ερωτήσεις ε, απευθύνθηκαν στον κλάδο των αυτοκινήτων. Το δικό μας το όραμα είναι ότι αυτά τα συστήματα, τα αυτόματα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, μπορούν να οδηγήσουν σε, σε μια νέα στροφή στην κινητικότητα. αυτό που μας είπε η κυρία Τελμόντε και σήμερα, ότι αυτά τα οχήματα μπορούν να έχουν τεράστιες ε, δυνατότητες αν θεωρήσουμε ότι πρόκειται για ένα νέο σύστημα. Δεν θα είναι ιδιοκτησία ενός αυτοκινήτου, αλλά θα είναι ε, ε, η υπηρεσία της κινητικότητας, ε, θα μοιράζεται κανείς αυτοκίνητο. Ε, γνωρίζουμε ότι αν πάμε προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορέσουν να γίνουν πολλές βελτιώσεις σε επίπεδο πόλεων. Εάν όμως πάνε τα πράγματα προς την άλλη κατεύθυνση, σίγουρα θα μπορέσουν να υπάρξουν κάποιοι πολύ σοβαροί κίνδυνοι. Γι' αυτό ακριβώς επικεντρωνόμαστε και στο αστικό επίπεδο. Αυτά τα συστήματα βέβαια δεν μπορούν να συνεισφέρουν μόνο σε αστικό επίπεδο, αλλά και στους αυτοκινητοδρόμους. Παραδείγματο χάρη οδηγούς ε, στον αυτοκινητόδρομο, το, ανθρώπους οι οποίοι οδηγούν για ώρες, ε, το να μπορούν να μείνουν στη λωρίδα τους είναι πολύ σημαντικό, να μην ε, χάνουν την προσοχή τους. Είναι πολύ σημαντικά λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα. Η έκθεσή μας δεν επικεντρώνεται σε ένα μόνο πράγμα. Ε, λέμε ότι μπορούμε να έχουμε διάφορες εφαρμογές προσαρμοσμένες στις ανάγκες. Αυτό το οποίο διευκρινίζουμε στην εκθεσή μας είναι ότι η πλήρης αυτοματοποίηση θα έρθει πολύ πιο μακροπρόθεσμα για αρκετούς λόγους και για λόγους ασφαλείας διότι ακόμα και οι δοκιμές ε, αυτών των ε, οχημάτων πρέπει να προσαρμοστούν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ε, δοκιμή η οποία θα μπορούσε να γίνει για να επιβεβαιώσει την ασφάλεια αυτών των μέσων. Ακόμα και στις Ηνωμένε Πολιτείε δεν υπάρχει, διότι αν παρακολουθήσετε τι γίνεται με τα αυτοκίνητα της Google, η Google αναγνωρίζει ότι μπορεί να υπάρχει ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό, ε, δεν χρειάζεται όχημα, χρειάζεται ένα μηχάνημα το οποίο αναγνωρίζεται ως οδηγός του οχήματος, αλλά η Google σαφέστατα είπε ότι ναι μεν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν δοκιμές ε, για να επιστοποιήσουν την απόδοση αυτού του οχήματος. Μάλλον όχι η Google, η εταιρεία, η επιχείρηση πιστοποίησης, η εταιρεία Μα ανησυχούν λιγότερο κάποιε άλλε πτυχέ και μα ανησυχούν λιγότερο γιατί πιστεύουμε ότι το νομικό πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή μπορεί ήδη να αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα, διότι θα κινηθούμε προς ένα σύστημα όπου ε, θα υπάρχει περισσότερο θέμα ευθύνης της κατασκευής του προϊόντος. Αλλά σίγουρα ο νομοθέτης θα πρέπει να εξετάσει ενδελεχώς τη διαδικασία και να δει και τι νομικά μέσα χρειάζονται, διότι σίγουρα κάποια πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν σε σχέση με την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τον ασφαλιστικό κλάδο, με τον οποίο μιλήσαμε κατά την εκπόνηση τη εκθεσή μα, ε, ε, και τους ρωτήσαμε αν αναμένουν μεγάλες απώλειες από ε, τη χρήση σε πιο, αυ... πιο αυτόνομων οχημάτων. Δεν πιστεύουν ότι θα υπάρχει κάτι τέτοιο. Διότι όπως σας είπα θα περάσουμε προς ένα σύστημα όπου θα υπάρχει ευθύνη της κατασκευής του προϊόντος. Επίσης σας είπα ότι το θέμα της αποδοχής από πλευράς ε, του κοινού είναι σημαντική. Πρέπει να το δούμε αυτό, διότι ακόμα έχουν επιφυλάξεις οι πολίτες για να χρησιμοποιήσουν τέτοιες τεχνολογίες. Ε, στο τέλος θα χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουν αυτά τα οχήματα καταναλωτές. Κάποιο αναφέρθηκε και σε μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή υπηρεσία για να ασχοληθεί με αυτές τις τεχνολογίες. Να σας πω ότι εάν ε, θέλουμε να δούμε αν ε, θα μπορέσει να υπάρξει διάθεση στην αγορά αυτών των οχημάτων, σκεφτείτε ότι θα χρειαστεί κάποιος διεθνής οργανισμός για να μπορέσει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Υπάρχει η Επιτροπή για την Ευρώπη, η οποία κάνει ουσιαστικό έργο, θα μπορούσε ίσως να αποτελέσει ε, το υπόβαθρο για να προχωρήσουν τα θέματα αυτά και να, τα, να δει και τις ανάγκες σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τώρα ο κύριος Νόγκεμπάμα. Ευχαριστώ. Πολλά θα μπορούσα να πω, αλλά θα περιοριστώ σε τεχνικές απαντήσεις που μπορώ να δώσω ως πρόεδρος του έτρα. Κύριε Φαντεκάμπ και κύριε Ρικέ, Είπατε ποιο είναι το χρονικό όριο. Μα το λέμε στην παρουσίασή μας. Αυτή τη στιγμή είμαστε ήδη στο επίπεδο 2, είναι οχήματα τα οποία μπορείτε να αγοράσετε. Και είναι στο όριο μεταξύ του επίπεδου 2 και 3. Άρα δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί διαρκεί τόσο πολύ. Στο παρελθόν δεν είχαμε καθόλου τους αισθητήρε και τους υπολογιστές που να έχουν υψηλή απόδοση ώστε να μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε για αυτές τις ε, λειτουργίες. Τώρα εφαρμόζουμε τα συστήματα βοήθειας προς τον οδηγό. Ξέρετε ε, ήδη όλοι το σύστημα ABS, ε, των φρένων. Και αυτό είναι ένα σύστημα βοήθειας προς τον οδηγό και τέτοια συστήματα αναπτύσσονται όλο και περισσότερο. Τι θα γίνει αμέσως ε, στην επόμενη χρονική ε, στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πρώτα απ' όλα θα υπάρξουν τέτοια συστήματα στην, ε, ε στις πόλεις. Είναι ανεπτυγμένα και τα συστήματα. Βέβαια η οδήγηση στο αυτοκινητόδρομο είναι πολύ απλούστερη από την οδήγηση σε μια πόλη με πεζούς, με Συγγνώμη, λοιπόν, το σωστό είναι ότι επειδή είναι απλούστερη η οδήγηση στου αυτοκινητοδρόμου, πρώτα θα εισαχθεί στου αυτοκινητοδρόμου. Γιατί χρειαζόμαστε εκεί την αναγκαία υποδομή, η οποία μετά σταδιακά θα πάει και στι πόλει. Κύριε Έρτογκ και Μπαχ, αναφερθήκατε στο ενδεχόμενο ατυχημάτων. Τα αυτοματοποιημένα οχήματα θα έχουν πολύ υψηλότερο επίπεδο ασφαλεία. Αλλά 100% δεν υπάρχει. Σίγουρα θα συνεχίσουν να προκύπτουν ατυχήματα που δεν θα μπορεί να τα αποφύγει ακόμη και ένα αυτοματοποιημένο όχημα. Ως ε, κλάδος φοβόμαστε λιγότερο τις τεχνικές βλάβες γιατί τα συστήματα αυτοπαρακολουθούνται και αν ε, διαπιστώσουν μία βλάβη κλείνουν αυτόματα και ε, ενημερώνουν ότι υπάρχει πρόβλημα με μία προειδοποίηση. Ξέρετε λοιπόν ότι για παράδειγμα αν κάποια συστήματα μπλοκαρίσματος δεν λειτουργούν σωστά σε παγωμένο δρόμο ε, αυτό διακόπτονται και ενημερώνουν τον οδηγό. Υπάρχει περιπτώσεις, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα οχήματα δεν θα μπορέσουν να αποφύγουν το ατύχημα γιατί είναι αναπόφευκτο. Ε, και τίθεται το ερώτημα ποιο θα φέρει την ευθύνη. Ε, πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα και εδώ χρειαζόμαστε και την βοήθεια του Κοινοβουλίου. Τέλος. δεν έχει να κάνει με το ποιος θα είναι το ε, θύμα. Αυτό δεν το βλέπουν οι αισθητήρες για το ποιος θα είναι το θύμα. Απλώς θα προσπαθήσουν να το αποφύγουν και αν δεν μπορούν να το αποφύγουν θα προσπαθήσουν να φρενάρουν όσο είναι δυνατόν ε, για να μειώσουν τις επιπτώσεις του ε, ατυχήματος και μετά θα γίνει ό,τι ατύχημα απομένει να γίνει. Εδώ χρειαζόμαστε λοιπόν την βοήθεια του νομοθέτη. Χρειαζόμαστε διαδικασίε για τεστ και για έλεγχο για ε, να πούμε ότι ναι, εφόσον έχουν γίνει αυτά τα τεστ, έχουμε φτάσει στο αναγκαίο επίπεδο για να μπορέσει να εισαχθεί στην αγορά. Και επαναλαμβάνω, τα οχήματα θα είναι πολύ ασφαλέστερα από τα σημερινά. Αλλά οπωσδήποτε θα παραμείνει ε, ένα υπόλοιπο κίνδυνο. Κύριε Λούνγκραν κάνατε μια έκκληση για την ε, ευχαρίστηση του να οδηγεί σε αυτοκίνητο. Δυστυχώ θα πρέπει σε ένα βαθμό να σα απογοητεύσω. Και σήμερα ακόμη, όταν οδηγείτε, αν έχετε αγοράσει ένα αυτοκίνητο, τα τελευταία 10 χρόνια ε, έχουν μια σειρά από ηλεκτρονικά συστήματα, συστήματα ελέγχου. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν περισσότερη δυνατότητα επεξεργασία δεδομένων από τα πρώτα διαστημόπλια που πήγαν στο φεγγάρι. Ε, είναι πιο αξιόπιστα λοιπόν τα αυτοκίνητα γιατί εμείς χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο τις δυνατότητες απόδοσης των συστημάτων πληροφορικής από ότι για παράδειγμα ο κλάδος της διασκέδασης. Τα αυτόματα συστήματα είναι πάντα μία επιλογή. Τα επόμενα χρόνια δεν θα κυδεμονεύουμε τον οδηγό αλλά θα είναι απλώς μια προσφορά εάν επιθυμεί να την αξιοποιήσει ο οδηγός για συγκεκριμένες καταστάσεις οδήγησης. Έχουμε τη δυνατότητα, αν αναγκαίο, να παρεύουμε για θέματα ασφάλειας. Κύριε Ντέλη, αναφερθήκατε στο θέμα ε, ανταλλαγής δεδομένων. Τεχνικά και σήμερα έχουμε ανταλλαγή δεδομένων και λειτουργεί μια χαρά. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα είναι σε πολιτικό επίπεδο. Ποια στοιχεία πρέπει να ανταλλάσσουμε και με ποιου. και πρέπει να γίνει μια σαφής ε, διάκριση. Ποια στοιχεία. Πρώτα απ' όλα έχουμε ε, στοιχεία για την ασφάλεια που θα πρέπει να μπορούν να αποσταλούν σε όλους το περιβάλλον. Και μετά υπάρχουν και στοιχεία πολύ υψηλού ιδιωτικού χαρακτήρα που δεν αφορούν κανένα. Και μετά υπάρχουν και στοιχεία που είναι ανάμεσα, που με ανωνυμοποιημένη μορφή θα μπορούσαν να ανταλλάσσονται, για παράδειγμα, για το πώς κυκλοφορία υπάρχει, πώς θα προκύψει, και στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να ε, κοινοποιούνται για λόγους ελέγχου της κυκλοφορίας εάν ο οδηγός το επιτρέψει. Άρα το ζήτημα δεν είναι αν μπορούμε να ε, κοινοποιούμε στοιχεία, αλλά θα πρέπει να πούμε ποια πρέπει πάντα, ποια πότε πότε και ποια ποτέ. Τέλος. Κύριε Μπαχ, Είπατε ε, θα υπάρχει ένα ε, μοντέλο αυτοκινήτου όπως το Airbus. Νομίζω ότι, ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία είναι ε, υπερήφανη για τα προϊόντα της και γι' αυτό εμένει στον ανταγωνισμό. Γι' αυτό θέλουμε να συνεχιστεί ο ανταγωνισμός σε τελευταία ανάλυση. Θέλουμε να εξακολουθήσουν να υπάρχουν διαφορετικές αυτοκινητοβιομηχανίες και να υπάρχουν συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών, μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά ε, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε στην, ε, στην πρώτη φάση ε, όπου για παράδειγμα και σε άλλες περιπτώσεις έχουμε συντάξει προγράμματα για κοινή έρευνα για να θέσουμε μερικές θεμελιώδεις παραμέτρους για να δημιουργήσουμε μια τεχνολογική πλατφόρμα για όλους αλλά μετά βέβαια πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός για να παραμείνει ανταγωνιστική η Ευρώπη και ευρύτερα στον κόσμο. Και για την κοινή χρήση οχημάτων και μοντέλων δεν είναι πάντα ίδια αυτά τα θέματα, αλλά την κοινή χρήση οχημάτων, το car sharing, το στηρίζουμε ήδη από τώρα και το προωθούμε για να μειωθεί η κυκλοφορία στις πόλεις. Είναι στόχος μας για να υπάρχει περισσότερη ενεργειακή αποδοτικότητα. Υποστηρίζουμε ενεργά το car sharing. Δεν είναι λοιπόν ε, κάτι το καινοτόμο αυτό αυτά τα οχήματα όλο και περισσότερο αξιοποιούνται και όσο καλύτερη είναι η αποδοσή τους, τόσο το καλύτερο. Δεν είναι καμία ε, καινούρια αποφασιστική τομή αυτή για τον κλάδο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Στη Βρέμη το car sharing, η κοινή χρήση, ε, ε, κάθε τέτοιο αυτοκίνητο αντικαθιστά 10 αυτοκίνητα που αποσύρονται από την κυκλοφορία. Έχει συνέπειε. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Μίλλορ για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Για τη Σιόν που ρώτησε ο κύριος Βαντεκάμπ. Γιατί αρχίσαμε από τη Σιόν. Κάπου έπρεπε να ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα σε μια μικρή πόλη, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να συνεννοηθούν ε, και να πιστούν οι άνθρωποι. Είναι λιγότεροι αυτοί που πρέπει να πείσει. Γιατί το μεγαλύτερο εμπόδιο σήμερα δεν είναι το τεχνικό, είναι να πείσει τους ενδιαφερομένους και τους αρμοδίους να σου δώσουν την άδεια. Και ίσως είναι πιο εύκολο αυτό στην Ελβετία από τις άλλα μέρη, γιατί κάνουμε παγκοσμίω το πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα για αυτόματες ε, ε, αστικές συγκοινωνίες σε κανονικούς δρόμους. Βεβαίως περιορίζεται στο Δήμο και στην πόλη της Ιών. Αν θέλετε να πάτε από εκεί στο Βερολίνο δεν γίνεται, αλλά μέσα στην πόλη κυκλοφορεί. Επίσης στη Ιών, ε, κάναμε αυτό το πείραμα γιατί θεωρήσαμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να αντικαταστήσουμε τα λεωφορεία μας, τα μετρό ε, και τα τραμ. Αλλά τις υπηρεσίες χαμηλής πυκνότητας που είναι on demand, δηλαδή ε, γι' αυτό είναι πιο εύκολο να το βρει κανείς στην Ήπεθρο ή σε κάποια μικρή πόλη. Ε, σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφαλείας, γιατί μάλλον έτσι, στα τεχνικά θέματα δεν μπήκα σε λεπτομέρειες για να το ξεκαθαρίσω. Ε, αυτό το λεωφορείο δεν έχει ούτε θέση οδηγού, ούτε τιμόνι, ούτε φρένα, ούτε τίποτα ε, που να μπορέσει κάποιος να ε, πιάσει το τιμόνι. Έχει ένα κουμπί μόνο που είναι το stop για να σταματήσει. Βεβαίως μπορείτε να πείτε ότι αυτό είναι επικίνδυνο, αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, ένας εξαιρετικός ε, να μειωθεί, ο κίνδυνο είναι να μειωθεί η ταχύτητα. Το λεωφορέκι λοιπόν αυτό κυκλοφορεί με ταχύτητα μόνο 20 χιλιόμετρων την ώρα. Για αστική συγκοινωνία αυτό είναι καλό από ταχύτητα. Βεβαίως ε, μπορεί να πηγαίνει και πιο γρήγορα, αλλά για λόγους ασφαλείας ξεκινήσαμε από τα 20. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται ποτέ αυτά να γίνουν 200 χιλιόμετρα την ώρα. Αλλά με χαμηλή ταχύτητα μειώνεται και ο κίνδυνος ε, αρκετά και το πρόβλημα για να πατήσω στα γαλλικά στον κύριο Χικέ, για να τιμήσω ε, και το γαλλόφωνο τμήμα της δεύτερης πατρίδας μου που μειοθέτησε, ε, χρονικός ορίζον. Πέρσι ή πρόπερσι, έχετε δίκιο, θα έλεγα ότι πρέπει να περιμένουμε μια εικοσαετία. Τώρα δεν είμαι τόσο σίγουρος πια. Σήμερα υπάρχουν ήδη τα οχήματα και για την συγκεκριμένη εφαρμογή εδώ μέσα μαζικής μεταφοράς που υπάρχει ένας διαχειριστής και τα ελέγχει όλα αυτά και ένα δρομολόγιο πιο περιορισμένο ε, υφίσταται αυτή η δυνατότητα. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για να ε, προχωρήσουμε πιο γρήγορα είναι ακριβώς η νομοθεσία. Δηλαδή οι άδειε, οι εγκρίσει στην ε, Ελβετία περιμένουμε την έγκριση τύπου από ε, το αρμόδιο κρατικό φορέα. Έχουμε την επόμενο συνάδελφο στο επόμενο πάνελ που θα αναφερθεί σε αυτό από τον συγκεκριμένο οργανισμό. Αλλά θα πρέπει κάπως όλες οι νομοθεσίες να προσαρμοστούν στα μέσα μας μεταφορά δεν τίθεται τόσο πολύ το θέμα της ευθύνη, γιατί ήδη από σήμερα είμαστε υπεύθυνοι για τα οχήματά μας και έχουμε συνηθίσει να εγγυόμεθα την ασφάλεια στου επιβάτε και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη αν κάτι πάει στραβά. Ανησυχούμε λιγότερο από ότι για ένα κανονικό όχημα, διότι ε, έχουμε μια δεκαριά κάμερες και με λιγότερα προβλήματα για να αποδείξουμε ε, ποιος έφταιγε αν ήταν το δικό μας όχημα ή κάποιος άλλος. Ένας τρίτος. Δεν είναι αυτό το βασικό εμπόδιο. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι χρειάζεται προσαρμογή της νομοθεσίας. Μετά τίθεται το θέμα των υποδομών και μπορώ να σας διαβεβαιώσω, αντίθετα με προηγούμενες εμπειρίες που ήταν μάλλον δαπανηρές, διότι πρόκειται για τηλεκατευθυνόμενα οχήματα, Τώρα πρόκειται για ε, αυτόνομη τεχνολογία, δηλαδή δεν χρειάζεται καμία υποδομή. Η μόνη υποδομή που χρειάζεται στον αυτοκινητόδρομο είναι κάπου να βάλεις μία πινακίδα, ε, ένα stop για να περιμένει εκεί, που δεν χρειάζεται ούτε αυτό όταν έχεις εφαρμογή στο smartphone ε, για να παραγγείλεις να έρθει το αυτοκίνητο. Δεν χρειάζεται καν η πινακίδα δηλαδή για τη στάση, ότι εδώ πρέπει να το περιμένεις να έρθει να σταματήσει είναι καινούργια τα οχήματα, λίγα σε αριθμό στη σειρά παραγωγής, ηλεκτροκίνητα, ε, στάνταρ ε, με λογισμικό διαχείριση, με αισθητήρε, δεν είναι τόσο ακριβά όμως. Και βεβαίως είναι πολύ πιο φθηνά. Αν δεν το χρησιμοποιεί, όπως ακούστηκε, ένας άνθρωπος μισή ώρα τη μέρα, ε, αλλά αν το μοιράζονται περισσότεροι ή μεταφέρει περισσότερους επιβάτες ε, με μια εφαρμογή, ακόμα και σαν μαζική συγκοινωνία. Και τέλος η αποδοχή. Μέχρι στιγμής, εμείς ήδη μεταφέρουμε επιβάτες, κόσμο. Και εσείς όταν παίρνετε το λεωφορείο ή το μετρό δεν οδηγείτε εσείς και σας κάνει αυτό. Δηλαδή, ξέρετε ότι είναι καλή οργάνωση και καλή διαχείριση. Ε, το ίδιο περιμένουμε και από τα οχήματα αυτά. Οι πρώτες αντιδράσεις είναι πάρα πολύ θετικές και μας χαροποιεί. Και χαίρεται και ο κόσμος που κυκλοφορεί με τέτοια οχήματα. Για να εξηγήσουμε τη λειτουργία υπάρχει κάποιος στην αρχή που συνοδεύει και εξηγεί, αλλά δεν οδηγεί, εξηγεί. Πώς να οδηγήσει, αφού είπαμε ότι δεν έχει ούτε τιμόνι, ούτε φρένο, ούτε τίποτα και ακόμα και οι δημοσιογράφοι ε, από όλο τον κόσμο που ήρθαν και δοκίμασαν του τελευταίους μήνες το όχημα αυτό είχαν μάλλον θετικές αντιδράσεις, πράγμα που με σανθερίνει για το μέλλον γιατί συχνά είναι η πιο δύσπιστοι και οι πιο επικρίτικη Και είμαστε αρκετά αισιόδοξοι και απόλυτα αισιόδοξοι για τη χρήση τέτοιων οχημάτων στι αστικές συγκοινωνίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνει εδώ το πρώτο πάνελ και η πρώτη συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσα, και πάμε στο δεύτερο. Θα σας παρακαλούσα να έρθετε να λάβετε τις θέσεις σας. I think we can continue. Λοιπόν, ε, να συνεχίσουμε. Παρακαλώ, καθίστε. Περάμε τώρα στο δεύτερο γύρο ομιλιών για τα ΕΦΗ, e, συστήματα μεταφορών και την τιμολόγηση της κινητικότητας πρώτος είναι ο κύριος Eric Sampson από το Πανεπιστήμιο του Newcastle και έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορεί να σας λέω και πράγματα που ξέρετε, αλλά οι μεταφορές είναι πολύπλοκες. Υπάρχουν ε, συνεχώς ε, ζήτηση για περισσότερα και εντάσεις, γιατί δεν έχεις τη ε, δυνατότητα να δώσεις αρκετά περισσότερο ώστε να καλύψεις τη ζήτηση και κάποιοι συζητούν ε, τη μείωση της ζήτησης και πρέπει να, κάποιοι άλλοι συζητούν να αυξήσουμε την ε, προσφορά και πάντα τελικά κατασκευάζουμε περισσότερες υποδομές. Τα ευφυή e συστήματα μεταφορών είναι ένας τρόπος να αυξήσουμε τη ζήτηση χωρίς να χρειαστεί να κατασκευάσουμε νέες υποδομές. Προέκυψαν από εξελίξεις οι οποίες έγιναν τη διάρκεια πολλών ετών και σας έχω αναφέρει τις ε, όπω όπως αποκαλώ. Αυτό μας βοήθησε να έχουμε αυτές τις ευφύ μεταφορές και υποφεληθήκαμε και από αυτές. Δεν θα επιστρέψω σε λεπτομέρειες, τις περισσότερες αναγνωρίζετε, αλλά θα ήθελα να σταθώ σε κάποιες ως πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα έξυπνα τηλέφωνα, υπολογιστέ και τηλέφωνα ξέρουμε ότι γίνονται όλο και πιο έξυπνα, αλλά τελικά είναι ε, συσκευές συλλογής δεδομένων. Η ανάπτυξη τη συλλογή δεδομένων μεταμορφώνει την αγορά και έχουμε συνεχή μετατόπιση από την ιδιοκτησία προϊόντων στην παροχή υπηρεσιών από αυτά. Αυτά τα τρία μαζί δίνουν νέες δυνατότητες, νέες ιδέες, νέες ε, διαδικασίες, όπως για παράδειγμα την παροχή Υπηρεσίας κινητικότητας. Ε, υπάρχει όλο ένα και μεγαλύτερος έλεγχος λογισμικού στον τομέα της αεροπορίας. Ξέρετε ότι τα σύγχρονα αεροπλάνα δεν τα πετούν πιλότοι γιατί θα είναι πολύ δύσκολη αυτή η διαδικασία. Κάποιες τάσεις έχουμε και στις υπόλοιπες μεταφορές, ε, αυτόματο ε, σύστημα πέδησης, ε, υποβοηθούμενο παρκάρισμα και το καθεξής. Και όλα αυτά τα συστήματα ε, αντιδρούν πολύ περισσότερο από έναν άνθρωπο ο αερόσακος, για παράδειγμα, θα βγει πολύ πιο γρήγορα από ότι θα καταλάβει ένας άνθρωπος ότι πρόκειται να συγκρουστεί με άλλο όχημα. Υπάρχουν ε, αρκετά σημαντικά πράγματα ε, τα, στα συστήματα. Μπορούμε να έχουμε τεχνολογία που είναι πιο αποτελεσματική, πιο αποδοτική, πιο ασφαλής, πιο οικολογική, ε, πολύ πιο ασφαλής από οποιοδήποτε άλλο μέσο μεταφοράς. Με ένα τέτοιο λοιπόν οπλοστάσιο ε, εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας από όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα, ε, ποιο είναι το πρόβλημα ε, με την τεχνολογία αυτή. Η σύντομη απάντηση είναι ότι δεν μας λείπουν και πολλά πράγματα. Χρειαζόμαστε καλύτερες βαταρίες για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για τη φόρτιση των αυτοκινήτων και χρειαζόμαστε και οικονομικά συστήματα φόρτισης εν κινήσει. Πρέπει να γίνουν πιο έξυπνες οι υποδομές. Ε, εάν είχαν έρθει οι ε, άνθρωποι του 18ου αιώνα εδώ σήμερα, θα διαπίστωναν ότι τα δικά δίκτυα δεν έχουν αλλάξει και πολύ από εκεί που τα άφησαν. Επομένως, χρειαζόμαστε κάτι το οποίο να είναι πάρα πολύ έξυπνο. Πρέπει να αναπτύξουμε διαδρόμους για πλήρως αυτοκινητωμένα, αυτοματοποιημένα αυτοκίνητα μέσω συνδεδεμένων αυτοκινήτων. Και επομένως πρέπει να έχουμε και καλύτερους και φθηνότερους αισθητήρε, πρέπει να έχουμε βελτίωση της τηλεφωνίας ε, για τα συστήματα αυτά, που σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί και επέκταση των δικτύων κινητή τηλεφωνίας. Αυτό έχει αναφερθεί ήδη. Κάποιοι άλλοι αναφέρθηκαν στην ε, διασύνδεση των οχημάτων και το γεγονός ότι πηγαίνουμε ε, στον περίεργο κόσμο του διαδικτύου των πραγμάτων, του Internet of Things και δεν γνωρίζουμε αρκετά και δεν κατανοούμε αρκετά για την κυβερνοασφάλεια αυτού του Internet των πραγμάτων. Αν πραγματικά λοιπόν θέλουμε να περάσουμε ε, επίσης και ως καύσιμο στο υδρογόνο, ε, πρέπει ε, να κάνουμε πολύ περισσότερα σε αυτό το τομέα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κατάλογο με διάφορες επιθυμίες και δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος αυτός ο κατάλογος. Εντός λίγο θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Τι άλλο μας λείπει λοιπόν είτε δεν αντιλαμβανόμαστε ή δεν ε, αποδεχόμαστε αυτά τα πράγματα που μας βλέπει στον κατάλογο. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για τη ζήτηση στις μελλοντικέ μεταφορές και πώς θα διαμορφωθεί και επομένως τι θα κάνει αυτό ε, και τι συνέπειες θα έχει και για τα φορολογικά εισοδήματα. Δεν κατανοούμε καλά την οδηγική συμπεριφορά, το γεγονός ότι μπορεί να χάσει την προσοχή του οδηγός, ε, και την ε, υπερφόρτωση. Επίσης, ε, για τις εκπομπές του αυτοκινήτου, ο κόσμος της αεροπορίας επίσης ε, γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει κοινό έλεγχος, τι σημαίνει να γνωρίζει ο πιλότος ή ο οδηγός τι πρέπει να κάνει και πώς γίνεται να εκχωρήσει τον έλεγχο αλλά και να ξαναανακτήσεις τον έλεγχο του οχήματος. Όλα αυτά τα συζητάμε στα αυτόνομα οχήματα και δεν έχουν γίνει απόλυτα κατανοητά. Δεν αντιλαμβανόμαστε επίση τις εκπομπέ ε, των οχημάτων στον πραγματικό κόσμο, σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και επίσης δεν κατανοούμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή αυτό, οχήματα τα οποία μπορούν να έχουν ωφέλη και μπορεί να είναι πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο φθηνά από τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό. Ε, υπάρχει και ε, ένα σχετικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον οποίο θα μπορούσα να σας παραπέμψω. Επίσης, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι συνέπειες έχουν τα υψηλά αυτοματοποιημένα οχήματα, δεν λέω αυτόνομα, τι συνέπειες μπορεί να έχουν για την κίνηση, για το παρκάρισμα, για την ασφάλεια και φυσικά και τους φόρους όπως σας είπα και προηγουμένως. Και ακόμα δεν καταλαβαίνουμε το ρόλο των drones στις μεταφορές. Υπάρχει ρόλος και αν ναι ποιος είναι αυτός. Ε, κάτι άλλο που λείπει δεν υπάρχουν ε, προδιαγραφές για τη χαρτογράφηση. Η χαρτογράφηση με την πιο γενική της έννοια, το τι ακριβώς γίνεται στο ευρύτερο περιβάλλον, όχι ένας διδιάστατος χάρτης, αλλά κάτι που πιο περίπλοκο. Χρειαζόμαστε επίσης δεδομένα για το κόστος ωφέλεια ε, της ε, χρήσης αυτής της τεχνολογίας. Χρειαζόμαστε να μας πούνε οι επιστήμονες τι έκαναν και πώς επωφελήθηκαν από αυτές τις υποδομές. Επίσης, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανών και των ε, διαχειριστών των υποδομών. Δεν θέλουν να συνομιλήσουν και είναι πολύ περίεργο γιατί ο ένας εξαρτάται από τον άλλον. Πολλοί αναφέρθηκαν επίσης ε, στο ποιος έχει την ευθύνη και στο κατάλληλο νομικό πλαίσιο για τα υψηλά στους αυτοματοποιημένα οχήματα. Ε, και επίσης έχουμε πολύ μικρή πείρα για μικρές, ε, μικρό αριθμό οχημάτων. 5% έχω βάλει εγώ εδώ που θα χρησιμοποιούνται και θα είναι υψηλής αυτοματοποίησης. Χρειαζόμαστε επίσης περισσότερες δοκιμές για οχήματα που μεταφέρουν εμπορεύματα και χρειαζόμαστε και μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική. Γιατί, Γιατί έχουμε ανταγωνισμό και υπάρχουν διάφορε επιχειρήσει που ανταγωνίζονται μία την άλλη. Και όπω επίση αναφέρθηκε, έχουμε κάποιε μεγάλε, κυρίω αμερικανικέ επιχειρήσει που θέλουν να διεισδύσουν σε αυτό το χώρο για να μπορέσουν να λάβουν πληροφορίε για το εμπόριο και να μην, δεν ε, θέλουν απλώ ε, να ωφελήσουν του ε, ε, τις μεταφορές και τις μεταφορές. Εγώ όταν ήμουν παιδί, να σας δώσω μια εικόνα, σε εναρμολογούσα ε, μοντέλα. Όταν παίρνεις ένα μοντελάκι, παίρνεις τα διάφορα μέρη, τα τμήματα που το αποτελεί και ένα σχέδιο. Και ε, ο κόσμο των ε, υψηλά αυτοματοποιημένων αυτοκινήτων είναι κάτι αντίστοιχο. Έχουμε τα διάφορα εξαρτήματα, δεν έχουμε ακόμα τι οδηγίε όμω και δεν έχουμε εικόνα. Εκεί πρέπει να δράσουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ο Τόμ Φέγκε που είναι αναλυτής για θέματα μεταφορών στο Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών, ITF. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Α, ωραία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας. Είμαι από το Αμβούργο που είναι πολύ αγγλόφιλη πόλη ε, της Χανσιατικής Λίγας, οπότε θα μιλήσω αγγλικά. Τι είναι το φόρο μας. Είμαι τμήμα του ΟΣΑ στο Παρίσι. Είμαστε μια ομάδα μελετών, think tank. Συμμετέχουν 58 κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη του ΟΣΑ και άλλες χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα, δίνουμε συμβουλές για θέματα πολιτικής στους Υπουργούς Μεταφορών μας. Για μια σειρά θέματα. Πρέπει να προετοιμαστούν ε, για διάφορα θέματα και εμείς τους ε, δίνουμε την ενημέρωση και έχουμε μια συνάντηση ε, κορυφής, μια γενική συνέλευση που φέτος θα γίνει στη Λιψία και θα αφορά, θα αφορά τις πράσινες μεταφορές. Επίσης εκπονούμε μελέτες και τις δημοσιεύουμε. Εδώ βλέπετε δύο παραδείγματα που έχουν να κάνουν με το ρόλο μας για τις μεταφορές του μέλλοντος. Θα τα αναφέρω παρακάτω. Αλλά να σας πω ποια θέματα θεωρούμε ότι είναι σημαντικά. Έχουμε εργαστεί για τα μεγάλα δεδομένα και τις μεταφορές. Έχουμε κάνει μια πρώτη μελέτη για να καθορίσουμε το πεδίο εφαρμογής. Είναι στο site μας. Αυτή η εργασία συνεχίζεται. Κάποια δουλειά που έχουμε κάνει για μερικά πιο επιμέρους θέματα θα δημοσιευθεί σύντομα και μια άλλη μελέτη αφορά μια αναβάθμιση των, Ευρωπα... των ε, αστικών συστημάτων κινητικότητας. Προσπαθούμε δηλαδή να διαμορφώσουμε ε, ένα όραμα για ένα μεγάλο αριθμό οχημάτων ε, τα οποία τα μοιράζονται και είναι οχήματα αυτοματοποιημένα σε αστικές περιοχές. Είναι λοιπόν ε, πολύ ενδιαφέρουσε αυτές τις δημοσιεύσεις του οργανισμού μας, ITF. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, με ποιο τρόπο τα δεδομένα τροφοδοτούν την οικονομία. Το είπε και ο Έρη η συλλογή πολλών στοιχείων, όλο και μεγαλύτερου όγκου στοιχείων από νέες πηγές συλλογής, ο τρόπος οντοπισμού των και τα επιχειρηματικά πρότυπα που εξελίσσονται μπορούν να δώσουν απαντήσεις για αυτούς που διαμορφώνουν την πολιτική και μπορούν να επιτρέψουν νέες μορφές ε, κίνης, κινητικότητας ή νέες ε, προσεγγίσεις, νέα πρότυπα για την ε, κινητικότητα και έτσι ε, τροφοδοτούμε και την οικονομία. Πολλά στοιχεία για τον τομέα των μεταφορών είναι γεωτοπικά στοιχεία, δηλαδή συλλέγονται όπως κινούμε και ζω και εργάζομαι. Άρα θα πρέπει να μεταδίδονται, να κοινοποιούνται αυτά τα στοιχεία, πώς θα πρέπει ορισμένα να είναι να περιορίζονται στην ιδιωτική μου σφαίρα και πώς θα προστατευτώ από την εγκληματικότητα και την εγκληματικότητα. Ποιες είναι οι βασικές ε, ιδέες για την κινητικότητα. Πρώτα απ' όλα εξετάζουμε τη συμμετοχική οικονομία που μάλλον είναι καλό πράγμα αλλά εξετάζουμε και ποιε τεχνολογίε και ποια συστήματα προκύπτουν, όπω το Uber από αυτή την συμμετοχική οικονομία. Ορισμένα από αυτά θεωρείται ότι δημιουργούν ε, προβλήματα στις παραδοσιακές ε, επιχειρήσεις του κλάδου αυτού. Παρενοχλούν τη λειτουργία τους και οι ρυθμιστικές αρχές ε, τρέχουν και δεν φτάνουν. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να τα εντάξουμε στην οικονομία μας, πρέπει το ρυθμιστικό πρότυπο να αλλάξει. Πώς θα επιτρέψουμε αυτά τα συστήματα να ε, μπουν σε ένα κανονιστικό πλαίσιο. Και τέλος, θέλω να σας μιλήσω για τα νέα πρότυπα ε, κοινή κινητικότητας, μοιρασμένη κινητικότητας. Θα μπορούσαν δηλαδή οι αυτοκινητοβιομηχανίες να παρέχουν κινητικότητα. Ήδη γίνεται αυτό. Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες διαχειρίζονται συστήματα ε, κοινή χρήση οχημάτων. Υπάρχουν και πολλά άλλα άτυπα τέτοια ε, προγράμματα κοινή χρήση οχημάτων, αλλά ορισμένα γίνονται όλο και πιο μη άτυπα γίνονται επιχειρήσεις όπως το Uber. Αλλά υπάρχουν προβλήματα λοιπόν. Πώς μπορούν να ενταχθούν στην οικονομία κάποιων χωρών, γιατί ορισμένε φορέ με πολύ επιθετικό τρόπο προσπαθούν να εισέλθουν στην αγορά. Έχουν όμω και πολλέ ε, θετικέ επιπτώσει. Για παράδειγμα, οι συμφορήσει στου δρόμου μα έχει να κάνει με το γεγονό ότι ο μέσο αριθμό επιβατών στα οχήματα είναι 1,2. Όλε αυτέ οι νέε μορφέ αυξάνουν αυτόν τον αριθμό. και θα σας μιλήσω για την αναβάθμιση των συστημάτων κινητικότητας της πόλης. Δηλαδή, αν δημιουργήσουμε ένα σύστημα κοινής χρήσης ε, αυτομάτων αστικών συστημάτων κινητικότητας. Εξετάσαμε δύο διαφορετικές λύσεις, δύο διαφορετικά συστήματα στη μελέτη μας. Μία είναι πιο πολύ σαν ταξί. Ένα μικρό όχημα που επιτρέπει όμως την κοινή χρήση θα πάτε από εκεί που θέλετε να πάτε στον προορισμό σας, αλλά κάθοδον, χωρίς ε, να χρειάζεται να κάνετε μεγάλες ε, παρεκβάσεις, θα μπουν και άλλοι ένα ή δύο μέσα στο αυτοκίνητο. Και το άλλο θα ήταν ένα μεγαλύτερο όχημα με 10-12, όπου θα έπρεπε να κάνουν λίγο μεγαλύτερες παρακάμψεις βέβαια για να τους ε, παραλάβουν όλους αυτούς και δεν θα ήταν πάντα από την πόρτα σα ε, εκεί ακριβώ που θέλετε να πάτε θα μπορεί να είναι από κάποια στάση σε κάποιο άλλο σημείο θα χρειαζόταν δηλαδή να περπατήσετε και κάποιε εκατοντάδε μέτρα να δούμε ποιε είναι οι επιπτώσει στην κινητικότητα όλα αυτά και με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να αποφύγουμε το 90% των οχημάτων που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στου ε, δρόμου. Αυξάνοντα λοιπόν ε, τον αριθμό ε, επιβατών αν αυτοκίνητο θα ελευθερώναμε ένα μεγάλο τμήμα του αστικού χώρου για άλλες χρήσεις. Αλλά, τι θα το θέμα. Ποιος θα μας χορηγήσει αυτά τα νέα οχήματα. Μπορεί η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία να συνεχίσει να λειτουργεί και να αντιμετωπίσει εξελίξεις όπως στην Καλιφόρνια για παράδειγμα βλέπουμε ότι ήδη ε, προσπαθούν ήδη να περάσουν από αυτοκινητοβιομηχανίες σε παρόχους ε, υπηρεσιών κινητικότητας και από το να είναι γενικά αυτοκινητοβιομηχανίες να γίνουν ε, βιομηχανίες που παράγουν ειδικευμένα οχήματα και υπηρεσίες κινητικότητας. Ποιος θα λειτουργεί λοιπόν αυτά τα συστήματα. Θα είναι αυτοκινητοβιομηχανίες θα μετατραπούν σε κάτι τέτοιο, σε παρόχους. Θα είναι οι παραδοσιακοί πάροχοι των υπηρεσιών συγκοινωνιών, λεωφορεία, υπογείους και τέτοια αυτοί ή θα προκύψουν εντελώς νέα εγχειρήματα, ίσως από άλλες περιοχές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά προσπαθούμε να εξετάσουμε για να δώσουμε συμβουλές στους υπουργούς μας ε, κατά τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Σεβάστηκα σχεδόν ε, τα 7 λεπτά. Είμαι λοιπόν σχεδόν αποτελεσματικός ως Γερμανός. Ευχαριστώ πολύ και για την τήρηση του χρόνου, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι αρχίσαμε αργότερα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θέμε όμως γι' αυτό. Επόμενος, ε, ο μιλητής είναι ο κ. Ραφαλ Κέσλι από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Τοπίας της ε, Ελβετίας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που έχω να σας παρουσιάσω την εκθεσή μας. Σύντομα. Το πρώτο ήταν η εντολή, οι ορισμοί και οι στόχοι του mobility pricing και διάφορα μοντέλα για το σιδηρόδρομο και τον αυτοκινητόδρομο. Σε περίπτωση που έχουμε χρόνο θα σας μιλήσω και για το τέλος ε, που καταβάλουν τα φορτηγά και το ITS. Ε, όπως μπορείτε να δείτε από τη διαφάνεια, αναλάβαμε ε, από την περασμένη θητεία ε, την εντολή και το αρμόδιο, περιβάλ, ε, το αρμόδιο τμήμα μάλλον του ε, οργανισμού μας ανέλαβε μέχρι τα τέλη του 2015 να κάνει αυτή τη μελέτη. Ποιο ήταν ο στόχος. Να δούμε ποιο είναι ακριβώς ο στόχο ε, της τιμολόγηση των διοδίων για τον αυτοκινητόδρομο, για το σιδηρόδρομο και να χρησιμοποιηθεί αυτό ως βάση για μια κοινωνική και οικονομική και πολιτική συζήτηση. Στόχος λοιπόν και ορισμοί. είναι τα διόδια που πρέπει κάποιος να καταβάλει όταν χρησιμοποιεί μια υποδομή, ε, είτε είσαι γεωταχή, είτε είσαι δημόσια συγκοινωνία, ε, για να έχει ως στόχο το να επηρεαστεί η ε, ζήτηση. Στόχος είναι να εξομαλυνθεί κάπως η κυκλοφορία και η χρήση των υποδομών. Ο στόχος δεν είναι πρακτικός δεν είναι ε, στόχος να συλλεγούν κάποια έσοδα, ακόμα και αν φαίνεται εκ πρώτης όψεως ε, ούτε είναι ο στόχος να προστατεύεται το περιβάλλον. Ε, η ρύθμιση της κυκλοφορίας είναι ο βασικός στόχος. Εδώ βλέπετε τα πέντε μοντέλα και τις δυνατότητες που έχουμε για τους αυτοκινητοδρόμους. Το χιλιομετρικό το, ε, και φαίνεται ήδη από την πρώτη ε, πρόταση, όταν έχουμε το δίκτυο Α ας πούμε, και ε, χρησιμοποιείται για τους αυτοκινητοδρόμους και μάλιστα είναι χιλιομετρική η καταβολή του τέλους. Σήμερα υπάρχει ένα σύστημα καταποκοπήν δηλαδή, και προχωρούμε προς ε, την κατεύθυνση pay as you δηλαδή ο καθένας να πληρώνει για τα χιλιόμετρα που διανύει. Αυτό ε, δεν προσφέρεται για να ρυθμίζεται η κυκλοφορία. Στο δίκτυο Β, ε, για τη χρήση του οδικού εθνικού δικτύου υπάρχει χιλιομετρική χρέωση αλλά και έξτρα χιλιομετρική χρέωση όταν είναι ώρες αιχμής. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος να πάνε από παρακαμπτήριους δρόμους ή παραδρόμους και να μεταφερθεί εκεί η συμφόρηση. Ε, την επόμενη ε, πρόταση, ε, ζώνη δίκτυο, ζώνη α. Και πάλι χιλιομετρική χρέωση με έξτρα ε, στις ώρες αιχμής. Αλλά ε, όχι μόνο στο εθνικό δίκτυο, αλλά και στο αστικό δίκτυο. Επόμενη πρόταση, ζώνη δίκτυο, ζώνη β. Η διαφορά με την προηγούμενη είναι εξή και μόνο. Ότι ε, καταβάλλεται ε, ένα δυο ανάλογα με την απόσταση, ε, τη χιλιομετρική, ανεξαρτήτως ώρας, είτε είναι ώρα είτε όχι. Και η τελευταία ε, πρόταση αφορά ε, όλους τους εθνικούς δρόμους, τους ε, περιφερειακούς, τους μικρούς και αγροτικούς και τους δρόμους μέσα στις πόλεις χρέωση και χιλιομετρική και έξτρα ανεξαρτήτως ορών εχμής λοιπά. Αυτό είναι μία αντιμετώπιση ενιαία για όλη την επικράτεια και έτσι αποσοβείται και ο κίνδυνος να φύγεις από ένα αυτοκινητόδρομο που έχει διόδια για να μεταφερθεί κυκλοφορία σε άλλο μικρότερο δρόμο. Να σας πω δύο λόγια τώρα για τις δημόσιες συγκοινωνίες. Ε, έχει σημασία να πούμε ότι η μεγάλη διαφορά ε, ανάμεσα των ε, δημοσίων και των ιδιωτικών συγκοινωνιών είναι ότι έχουμε εταιρείε μεταφοράς επιβατών ως επιπλέον παίκτη. Και υπάρχει και ένα σύστημα flat rate που είναι ε, μία κάρτα απεριορίστων διαδρομών που μπορεί να χρησιμοποιεί ο επιβάτης, ε, πράγμα που δεν γίνεται στον αυτοκινητόδρομο. Βλέπετε εδώ τις τρεις ε, επιλογές και εκδοχές που έχουμε για τις δημόσιες συγκοινωνίες. Όταν έχουμε λεωφορεία, τρένα ή τραμ ε, που έχουν μεγάλη ζήτηση πληρώνουν οι επιβάτες ανάλογα με το χρόνο και με τον τόπο. Ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι σκόπιμο να διαφέρει και το εισιτήριο ανάλογα με τη ζήτηση και την ώρα αιχμής ή όχι. Βέβαια, μια τέτοια λύση είναι μόνο πιλωτική και δεν μπορεί κανείς να τη θεωρεί βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Δεύτερη πρόταση. Αυτό δεν εφαρμόζεται μόνο σε συγκεκριμένες ε, γραμμές, σε δρομολόγια, αλλά και σε συγκεκριμένες περιοχές ε, και σε διαφορετικό χρόνο και στο δίκτυο που αντιστοιχεί σε όλη την επικράτεια στον αυτοκινητόδρομο. Δεν αφορά αυτό μια συγκεκριμένη πόλη, μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά το σύνολο της χώρας σε όλη την Ελβετία. Ε, pay as you use, δηλαδή ο καθένας ε, πληρώνει ό,τι χρησιμοποιεί ποιοτικά και χρονικά. Για να υπάρχει μια πιο ομοιόμορφη κατανομή, ο καθένας πληρώνει, λοιπόν, ανάλογα με την υπηρεσία που χρησιμοποιεί. Έχω μερικά δευτερόλεπτα για να σας πω δύο λόγια. Ήδη σήμερα έχουμε τιμολόγηση της κινητικότητας ε, όταν υπάρχει βαριά κυκλοφορία. Ε, ε, των βαρέων οχημάτων δηλαδή. Το ITS που είναι τα FEE συστήματα μεταφορών συνδυάζεται η ευφυής κινητικότητα και αλλάζει την σημερινή ριζικά. Και θα πρέπει το κράτος να ε, κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή και να την ενισχύσει. Σας παραπέμπω στην ιστοσελίδα μας, αν θέλετε περισσότερα. Εκεί έχετε σε τρεις γλώσσες την έκθεση ε, και μπορείτε να τρέξετε σε περισσότερες ε, λεπτομέρειες. Ευχαριστώ κύριε Κέσλι. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Εύα Σόφκα, συντονίστρια του προγράμματος του Ινστιτούτου της Βαρσοβίας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι. Κύριε Πρόεδρε, είμαι από το Ερευνητικό Ινστιτούτο για Όδους και Γέφυρες που εδρεύει στη Βαρσοβία και θα ήθελα να σας πω που επικεντρώνεται η εφαρμοσμένη έρευνα. Θα είναι σύντομη η παρουσίαση και ελπίζω να μπορέσουμε να το συζητήσουμε αργότερα αν έχετε ερωτήσεις. Καταρχάς θα ήθελα να σας δώσω μια σύντομη εικόνα επιλεγμένων τεχνολογιών για την κινητικότητα. Θα μιλήσω για τα FEE συστήματα μεταφορών, το ITS και την κινητικότητα. Συμμετέχουμε ως Ερευνητικό Ινστιτούτο σε ένα από τα προγράμματα του Ορίζοντα 2020 ε, και ε, πρόγραμμα το οποίο έχει ε, χρήστες υποδομών, χρήστες γενικότερα σε όλα τα μέσα. Δεν αναφέρεται μόνο στα οδικά δίκτυα που είναι πολύ σημαντικά τη σήμερον ημέρα, αλλά αναζητούμε και τεχνολογίες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και σε άλλα μέσα μεταφοράς. Έχουμε λοιπόν ολοκληρωμένες υποδομές μεταφορών, συστήματα πληροφοριών, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα αυτή τη στιγμή και μας δίνει και ένα κατάλληλο περιβάλλον για να μοιραζόμαστε πληροφορίες για ευφυή συστήματα, για διόδια, για κινητικότητα χρηστών και για αυτοματοποίηση. Κάτι άλλο το οποίο θέλω να σας δείξω, ε, που είναι τμήμα του προγράμματός μας, είναι η αυτοματοποίηση. Το προηγούμενο πάνελ αναφέρθηκε στα ε, αυτοκινούμενα οχήματα, εγώ θα ήθελα να σταθώ στην επικοινωνία, που είναι πολύ σημαντικό τμήμα τη τεχνολογία που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή και θα είναι και στο μέλλον. Υπάρχει επικοινωνία από όχημα σε όχημα, από όχημα σε υποδομή και όχημα και υποδομή προ το χ, που είναι διάφορε συσκευέ ή διάφορα ανέφη πληροφοριών τα οποία μεταβιβάζονται μέσω του ίντερνετ των πραγμάτων. Επίσης, ως Ερευνητικό Ινστιτούτο, πρόσφατα ξεκινήσαμε και μια συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Συστημάτων Μεταφορών που εδρεύει στην Τσεχία ε, και κυρίως συλλέγουν ε, big data. Τι είναι αυτά τα big data, τα συζητούν όλοι. Πρόκειται για ένα τεράστιο αριθμό δεδομένων τα οποία δημιουργούνται και δημιουργούνται και από διάφορα μέσα μεταφοράς, ε, καθώς επίσης και από διάφορα τμήματα της μεταφοράς, ακόμα και από ε, την αυτοματοποίηση και τον κλάδο των ιδιοκτήτων των οχημάτων. Σε ποιον ανήκουν αυτά τα δεδομένα είναι το μεγάλο ερώτημα και κατά πόσο μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, ώστε να μπορέσουν να ε, λειτουργήσουν και εποφελεί των χρηστών. Αυτά είναι τα βασικότερα προγράμματα στα οποία ε, επικεντρωνόμαστε και θα δούμε πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για μας, για τους πελάτες, ώστε να έχουμε βελτιώσει στη μεταφορά και ε, στους τρόπους μεταφοράς. Big data λοιπόν για την κινητικότητα και την κίνηση. Αν μπορούμε να το μετρήσουμε, τότε δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε μοντέλο γι' αυτό. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ερωτήματα, είναι ένα από τα θέματα που θέλουμε να προωθήσουμε στην έρευνά μας, ε, αλλά και σε εσά διότι είναι πολύ πιο εύκολο να μετρήσουμε κάτι χωρίς να χρειαζόμαστε ένα μοντέλο για να το μετρήσουμε. Και η σημερινή τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να μετρήσουμε με μεγάλη ακρίβεια την κίνηση και να τη διαβιβάσουμε στους τελικούς χρήστες, δηλαδή εμάς, τους οδηγούς, τους ανθρώπους που διαχειρίζονται τα, οδικά, τα οδικά δίκτυα, δίκτυα επιμελητίας επίσης και όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτοματοποίησης που διαθέτουν τα οχήματα ήδη. Δυστυχώ, ε, δεν έχω τη δυνατότητα να σα παίξω το βιντεάκι εδώ. Είναι ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Είναι ένα όχημα το οποίο οδηγεί. Υπάρχουν αισθητήρε παντού, επομένω μπορούμε να δούμε τη σηματοδότηση, ε, διάφορα στοιχεία τα οποία μα δείχνουν τα ωραία ταχύτητα, ε, πληροφορίε για τον ταξιδιώτη, για το τον καιρό και οτιδήποτε σημεία συμφόρησης και όλα αυτά μπορούν να τα δώσουν και μέσω του GPS αλλά και άλλων συσκευών που μπορούν να μας δώσουν στοιχεία όπως οδηγούμε. Αυτά τη στιγμή αυτά διατίθενται ήδη αλλά σε ένα αυτοματοποιημένο όχημα θα μπορούμε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια ε, και να υπάρχει και επικοινωνία μεταξύ των οχημάτων και μεταξύ του οχήματος και της επιδομής και να βελτιωθεί κιόλας. Επίσης, θα ήθελα να σας δείξω και αυτή την ανάλυση εθνικής κινητικότητας που γίνεται στην Τσεχική Δημοκρατία βασίζεται σε σύνολα ε, για την, το σημείο καταγωγής, το σημείο προέλευσης και το σημείο προορισμού. Εδώ έχουμε τους αστερίξους που δείχνουν ε, τα διάφορα σημεία και εδώ βλέπουμε πώς αντικατοπτρίζονται σε πραγματικό χρόνο ε, τα, που βρίσκεται κάποιος, αν πηγαίνει από το, ένα σημείο στο άλλο και ούτω καθεξής. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σήμερα. Ε, διατίθεται από την ιστοσελίδα Ρόντος και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί μπορούμε να δούμε πώς πραγματικά ε, υπάρχει κινητικότητα σε πραγματικό χρόνο και υπάρχει και ο Άτλας για την κεντρική ευρωπαϊκή κινητικότητα. Τα κόκκινα σημεία είναι τα σημεία ε, συμφόρησης ε, και τα σημεία συγκέντρωσης κινητικότητας. Αυτά τα στοιχεία είναι διαθέσιμα διαδικτυακά και μπορούν να χρησιμοποιούν για διάφορους ε, σκοπούς, κυρίως για τη διαχείριση της κίνησης, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους λόγους, για εμπορικούς σκοπούς, για ηλεκτρονικό εμπόριο, για μεταφορά ανθρώπων και αγαθών, για θέματα εφοδιαστική επιμελητία. Αν μπορούμε να έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία, μπορείς να προγραμματίσεις και το μέλλον του πώς θα μεταφέρεις τα πάντα. Κάποιες από τις εφαρμογές οι οποίες είναι διαθέσιμες χρησιμοποιώντας ε, Big Data και τα στοιχεία που λαμβάνουμε από του αισθητήρε είναι στοιχεία για τη διαχείριση της κίνησης μέσω του ρόντος. Αυτό είναι διαθέσιμο ε, στους υπολογιστές ε, ή και στα Palm Top και στους, ε, στα GPS μπορεί ο καθένας να δει χάρτες κίνησης. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό προϊόν. Πρόκειται για μια εφαρμογή που βοηθά τα κέντρα διαχείρισης κίνησης να διαχειρίζονται την κίνηση. Και εμείς ως χρήστες μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία αυτά στα οχήματά μας. Επίσης, εδώ έχουμε παρακολούθηση της κίνησης της Σλοβακίας βάσει GPS. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για διαχείριση εκδηλώσεων. Ε, επειδή είναι μεγάλη αβεβαιότητα στη ζωή μας σήμερα, διότι δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αλλάζει το κλίμα, έχουμε τρομοκρατικές επιθέσεις και πρέπει κάπως να διαχειριστούμε διάφορες μεγάλες εκδηλώσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε να συμβεί κάτι και έχουμε εμεί οργανώσει μια εκδήλωση. Αυτό ε, το σύστημα μας δίνει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, πώς μπορείς να κατευθύνεις προς άλλη κατεύθυνση τους ε, ανθρώπους, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι πολύ καλό εργαλείο. Και τέλος έχουμε ε, διαχείριση της κίνησης από άλλες πηγές. Μπορούμε να έχουμε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, για παράδειγμα, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. και στη διάρκεια της εκδήλωσης υπάρχει μια εφαρμογή που θα μπορούσε ε, να εστιάσει απευθείας μέσω Zoom ε, στην εκδήλωση για να δει τι συμβαίνει ε, και να αλλάξει τα πράγματα. συζητούμε λίγο και το θέμα της ε, ηλεκτρονικής ετικέτας και της κυκλοφοριακής συμφέρεσης. Το συζήτημα αυτό είναι και πολύ πολιτικό βέβαια, αλλά εγώ θα ήθελα να σας πω δύο λόγια. Αυτή τη στιγμή στην Πολωνία έχουμε ένα ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων για τα βαρέα οχήματα και αυτό γίνεται μέσω μιας συσκευής ε, που βρίσκεται εντός του οχήματος. Και έχω και ένα πολύ ωραίο διάγραμμα, το οποίο δυστυχώς ε, δεν ε, το βλέπετε, γιατί σε αυτόν τον υπολογιστή δεν έχετε αυτές τις λειτουργίες. Υπάρχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα λοιπόν διοδίων. Προσπαθούμε να έχουμε ένα ενοποιωμένο σύστημα συλλογή των δεδομένων και φυσικά η διαλειτουργικότητα είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ έχουμε τα στοιχεία του χρήστου, χρήστη, ε, μπορούμε να δούμε τι γίνεται με τη ροή, μπορεί να γίνει μεμονωμένα, ε, να το δούμε για ένα χρήστη, αλλά μπορούμε να το δούμε και από πλευράς παρόχου. Εκεί έχουμε διαδικασίες διαλειτουργικότητας, οι διαδικασίες προχωρούν, υπάρχει και συμφωνία σε επίπεδο υπηρεσίας και βλέπουμε και τι γίνεται με την ανασφάλεια σε επίπεδο τιμών. Ε, και εδώ βλέπετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Έχουμε ένα ε, βαρύ όχημα το οποίο πηγαίνει στο ε, σταθμό συλλογής, αυτά γίνονται ηλεκτρονικά. Μετά γίνεται καταγραφία, ε, λαμβάνεται φωτογραφία, περνάει το όχημα, γίνεται καταγραφή των διοδίων και μετά γίνεται ταξινόμηση του οχήματος και συλλογή, πληρωμή δηλαδή των διοδίων, όλα αυτά ηλεκτρονικά χωρίς να πρέπει να διακόψει καθόλου την κίνησή του. Υπάρχουν φυσικά θετικά και αρνητικά στοιχεία τώρα για την τιμολόγηση ε, ε της κίνησης. Ε, έχουμε στοιχεία για το πώς ε, δέχεται ο κόσμος την τιμολόγηση και τη χρέωση των διοδίων. Υπάρχουν κάποια θέματα για τη χρήση δημοσίων υποδομών, αλλά σε γενικές γραμμές ο κόσμος είναι αντίθετος και να σας δείξω και γιατί. Έγινε μια έρευνα από κάποια Ινστιτούτα στην Ισπανία το 2014 και θα ήθελα να σας δείξω εν συντομία κάποια αποτελέσματα. Ένα 36% όσων απάντησαν είπαν ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται διόδια για μείωση της ρήπανσης ε, και κίνηση, δηλαδή να βασίζεται στα διόδια βάσει των χιλιομετρικής απόστασης που διανύεται. Αυτή είναι καλή ιδέα. Επίσης, εισοδήματα από τα διόδια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των υποδομών, είπε το 29% και ένα 33% είπε ότι είναι για να βελτιωθεί το, δικτό, το οδικό δίκτυο και οι υποδομές και οι δύο τελευταίε διαφάνειες. Ξέρω ότι έχω περάσει λίγο το χρόνο μου, αλλά ήθελα να σας δείξω λίγο την πολιτική στα γρήγορα. Ένα 80% είπε ότι τα όρια ταχύτητας θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται αντί των διοδίων, ένα 37% δεν είχε τίποτα να πει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας ω ερευνητέ, το γεγονό ότι κανεί δεν έχει ιδέα για το τι κάνουν αυτέ οι πολιτικέ και δεν έχουν καμία ιδέα για το τι γίνεται με τα διόδια. Ένα 39% λέει ότι ήδη πολλά πληρώνουν, Επομένω δεν χρειάζεται να υπάρχει και διαφορετικό τρόπο ε, τιμολόγηση. Ε, ε, ε, είναι απλώς πρόσχημα για να τους, εφαρμόσουν, να τους επιβάλλουν ε, και άλλα διόδια. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία παρουσίαση. Κλέρ Ντουπρέ, της Γενικής Διεύθυνσης ΜΟΥΒΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που είμαι τελευταία. Γιατί πολλές φορές υπερβαίνω το χρόνο μου, οπότε τώρα είμαι πιεσμένη. θα ήθελα να σας μιλήσω για την πλατφόρμα C-Pavla C-ITS. Μιλήσαμε για κοινή χρήση οχημάτων, αλλά δεν μιλήσαμε για τα συνεταιρικά οχήματα. Και λέω οχήματα, όχι αυτοκίνητα. Τα συνεταιρικά ή συνεταιριστικά οχήματα είναι οχήματα που όχι απλώς επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων, αλλά και με άλλους χρήστες ε, της οδικής υποδομής με, για παράδειγμα, μοτοσυκλέτες, αλλά ανταλλάσσουν μηνύματα και με την υποδομή. Την υποδομή που είναι αρμόδια για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Έχουμε κάνει πολλά το τελευταίο χρόνο γι' αυτό. Και εδώ είναι τουλάχιστον ε, τρεις συνάδελφοι που έχουν συνεργαστεί στενά μαζί μας, συμπεριλαμβανομένου και του ΕΡΙΚ. Η συζήτηση έγινε μεταξύ ε, εμπειρογνωμόνων. Ε, ελπίζω να μπορούμε να θεωρηθούμε εμπειρογνώμονες. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι απόλυτα αναγκαίο, όχι μόνο μεταξύ εμπειρογνωμόνων, αλλά και για να ενημερώσουμε τους πολιτικούς. Και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στην Ολλανδική Προεδρία, γιατί είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί τους. Είναι σημαντικό οι δημόσιες αρχές που διαχειρίζονται τη μεταφορά, τις ε, μεταφορές να ξέρουν ποια είναι τα θέματα, να ξέρουν τι συζητάμε, να ξέρουν τι προκύπτει, αλλά να έχουν και τη δυνατότητα να προσανατολίσουν ε, την κατεύθυνση της καινοτομίας. Αναφερθήκαμε σε προθεσμίες 10 ε, χρόνια, 20 χρόνια, συνεργατικά συστήματα. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψω πώς θα συμβεί. Αλλά θα συμβεί οπωσδήποτε. Αλλά πώ ακριβώ είναι πολύ πιο δύσκολο να προβλέψω. Η ψηφοποίηση αλλάζει όμως τα πάντα. Αυτό το ξέρουμε. Συζητήσαμε για το ρόλο των δεδομένων για τα πολυτροπικά συστήματα. Το ίδιο ισχύει και για αυτό το θέμα που συζητάμε. Θέλουμε η καινοτομία να μας δώσει τις δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε τους στόχους μας, ε, συμφόρηση, οδική ασφάλεια και πρέπει να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ του κλάδου, των δημοσίων αρχών, των ερευνητών, των πολιτικών για να συμφωνήσουμε τι υπηρεσίες θέλουμε να μας παράσχουν αυτές οι τεχνολογίες. Βεβαίως είναι ζωτική σημασία σε όλα αυτά. Υπάρχουν και πολλές άλλες πρωτοβουλίες σε άλλα μέρη του κόσμου. Αλλά εμείς ως Ευρώπη δεν τα πάμε και τόσο άσχημα. Ορισμένες ε, επιχειρήσεις μας είναι πολύ ε, πρωτοπόρες σε κάποιο τομέα, άλλες σε άλλον, αλλά μας λείπει μια κεντρική προσέγγιση. Τι θέλουμε να επιτύχουμε, υπό ποιες συνθήκες και πότε. Γι' αυτό δημιουργήσαμε αυτή την πλατφόρμα που έχει θεωρηθεί πιστεύω πολύ λειτουργικό βοήθημα για να αναπτύξουμε αυτά τα συστήματα παντού στην Ευρώπη. Θα έλεγα λοιπόν ότι τον τελευταίο χρόνο που κάναμε πολλή δουλειά έχουμε τώρα μια ημερομηνία. Ο κλάδος μας έχει δώσει μια ημερομηνία. Όχι μόνο η αυτοκινητοβιομηχανία επιμένω. Είπαν λοιπόν ότι μέχρι το 2019 θα είναι έτοιμοι για να αναπτύξουν αυτές τις τεχνολογίες. Αλλά υπάρχουν πολλά θέματα. Και δεν είναι μόνο τεχνικά. Είναι πιο πολύ θέματα κοινωνικά, κοινωνίας. Για παράδειγμα, κύριε Ερτούγ, είπατε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα προστασίας των δεδομένων. Μα υπάρχει ήδη πλαίσιο που εγκρίθηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα από το Κοινοβούλιο. Αλλά βέβαια το να ξέρεις ποιες είναι οι αρχές είναι ένα θέμα. Το άλλο είναι πώς ε, στην πράξη θα εφαρμοστούν αυτές οι αρχές, τι λειτουργικές απαιτήσεις θα απορρέουν. Για παράδειγμα, είμαι στο αυτοκίνητό μου. Μιλήσαμε για διάφορα δεδομένα. Κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου ένα συνδεδεμένο και συνεργατικό αυτοκίνητο θα αποστέλει δεδομένα. Αλλά δεν είναι θέμα να πούμε ναι σε αυτά, όχι στα άλλα θα αποστέλλονται όλα αυτά τα δεδομένα συνέχεια. Θα πρέπει οι οδηγοί να είναι σε θέση να μπορούν να εκφραστούν και να πούν θέλω να ξέρουν που είμαι. Θέλω ε, να ενημερωθούν ορισμένες υπηρεσίες για το που είμαι ή όχι. Ο, η Επίτροπος Μπούλτς είπε πρόσφατα ότι τα στοιχεία για τον κλάδο δεν είναι τόσο θετικά. Είναι δεύτερη φορά, δεύτερη χρονιά που το λέει αυτό. Άρα το βασικό είναι να εστιάσουμε στις υπηρεσίες που θα ενισχύσουν την οδική ασφάλεια και που είναι εκατοντάδες. Χρειάστηκε να συμφωνήσουμε επί άνω των 100 συμμετεχόντων από τον κλάδο, τοπικές αρχές, ε, εθνικές αρχές, πάροχοι υπηρεσιών, τι, με όλους αυτούς αποφασίσαμε να συμφωνήσουμε σε ένα κατάλογο του τι υπηρεσίες θέλουμε. Και συμφωνήσαμε σε λίγο πάνω από 10 κατηγορίες εφαρμογών. Για παράδειγμα, έχετε μπροστά σας συμφόρηση, ορισμένα οχήματα κινούνται αργά. Θα μπορούσα να σας πω πολλά. Αλλά για να καταλάβετε ότι προσπαθούμε να συνδέσουμε το στόχο με την εφαρμογή του. Αναφερθήκαμε στην αυτοματοποίηση. Από την πλευρά μου, όπως είδατε και από το διάγραμμα του συναδέλφου από το τμήμα έρευνας, τα συνεργατικά συστήματα και η αυτοματοποίηση πρέπει να συμβαδίζουν. Και συνδυασμένα μπορούν να μας προσφέρουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, άρα δεν αντιπαρατίθενται. Και σίγουρα μόνη η αυτοματοποίηση δεν θα επιτύχει τους στόχους μας. Και γιατί όχι μόνη της. Για δύο λόγους. Νομίζω ότι η κυρία Ντεμόντε αναφέρθηκε στις αεροπορικές μεταφορές. Αν είσαι επιβάτης σε αεροπλάνο, αυτό που θες να ξέρεις είναι ότι το αεροπλάνο σου μπορεί να επικοινωνήσει με τον πύργο ελέγχου. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και με ένα αυτοματοποιημένο όχημα. Αλλά τώρα σε σχέση με την κίνηση. Τα οχήματα κυκλοφορούν σε δρόμους. Και οι δρόμοι έχουν κανόνες, όχι ευρωπαϊκούς, αλλά κανόνες που έχουν καθοριστεί από αυτούς που είναι αρμόδιοι για την κυκλοφορία τοπικά και εθνικά. Κανόνες για το πώς λειτουργεί το σύστημα των οδικών μεταφορών. Πρέπει λοιπόν όλοι όσοι εμπλέκονται ε, να μπορούν να έχουν το λόγο τους γι' αυτό. Αν θες για παράδειγμα να πεις ότι προσοχή εδώ σε αυτή την περιοχή υπάρχει ένα σχολείο, πρέπει να μπορείς να ε, ενημερώσεις γι' αυτό. Να το λάβουν όλοι υπόψη. Ποια είναι τα αποτελέσματα της εργασίας μας. Πρώτα απ' όλα καθορίσαμε μια σειρά από εφαρμογές που θεωρούμε ότι παρέχουν υπηρεσίες που θα πρέπει να εισαχθούν πρώτα. Ο στόχος είναι το 2019 να έχουν εισαχθεί αυτές οι υπηρεσίες. Επίσης έχουμε εργαστεί για θέματα διαλειτουργικότητα. Τα αναφέρατε και προηγουμένω όταν μιλήσατε για την αυτοματοποίηση. Γιατί δεν διασχίζουν μόνο τα οχήματα τα σύνορα. Ε, κάθε είδους ε, οχήματα ε, διασχίζουν σύνορα, άρα πρέπει να μπορούν να επικοινωνήσουν. Συζητήσαμε για τα τηλέφωνα. Όταν ε, χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σας δεν σας ενδιαφέρει ε, αν χρησιμοποιείτε Wi-Fi ή το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Θέλετε απλώς να επικοινωνήσετε. Το ίδιο θα πρέπει να είναι και για τα συνεργατικά συστήματα. Θα πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις υπάρχουσες τεχνολογίες. Να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις νέες μορφές και επίπεδα. Ελπίζουμε να αναπτυχθεί σύντομα και να ε, αναπτυχθεί παντού το 5G, το 5G. Αλλά ήδη να αξιοποιήσουμε αυτό που υπάρχει τώρα. Η έκθεση αυτή εγκρίθηκε ομόφωνα τέλος Ιανουαρίου. Πριν από μερικούς μήνες συμμετείχα σε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και να πω ότι ήδη το κείμενο αυτό, την έκθεση, την έχουν κατεβάσει 3.500 άτομα. Δεν είναι και άσχημα για έκθεση της Επιτροπής. Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Ετοιμάζουμε ένα βασικό πρόγραμμα, Master Plan, για την ε, περαιτέρω εισαγωγή του CITS ε, το τρίτο τρίμηνο και κάτι ακόμη. Είπατε πόσα έχουμε ως χρηματοδοτήσεις στο ε, ορίζον 2020 και το συγκρίνατε με τις χρηματοδοτήσεις της ΗΠΑ. Θα ήθελα να σας πω, μην εξετάζετε ένα συγκεκριμένο όργανο. Δείτε συνολικά τον ορίζοντα 2020. Δείτε και το CEF, ήταν νομίζω 70 εκατομμύρια για το CITS στο γενικό πακέτο χρηματοδότησης, στο γενικό πλαίσιο χρηματοδότησης. Και άλλες χρηματοδοτήσεις ήταν στα πλαίσια του συνολικού πλαισίου συνοχής. Αλλά ε, υπάρχουν και επιπλέον χρηματοδοτήσεις από τα κράτη-μέλη. Άρα δεν είναι και τόσο άσχημα τα πράγματα. Τέλος. Συνεργαζόμεθα με τον κλάδο, με τα κράτη-μέλη, για να υπάρξει μια κατεξοδότηση πράξη για το CITS. Είμαστε ακόμη σε πρώιμο αλλά θα επανέλθω όταν ε, έχουμε προχωρήσει λίγο παραπέρα για να σας ενημερώσω για το πώς πάει η κατεύθυνση την κατάλληλη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκαν εδώ οι παρουσιάσεις. Τώρα μπορούν να γίνουν και ερωτήσεις. Είμαστε σε πιο στενό κύκλο, αλλά δεν πειράζει. Βίμ Φαντακάμπ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ειλικρινά πρέπει να σας πω ότι... Πώς να το πω... Με έχουν κατακλείσει όλα αυτά τα δεδομένα, οι δυνατότητες, οι πληροφορίες. Ε, όλα αυτά, 9 η ώρα ξεκινήσαμε και ακόμα εδώ είμαστε. Ε, έχουμε γεμίσει πληροφορίες. Έχω τις εξής ερωτήσεις. Πρώτα στον κύριο Σαμσούν. Γιατί δεν έχουμε ακόμα μικρά ε, ηλεκτρο... ηλεκτρικές μπαταρίες ε, στοιχεία. Αυτό είναι θέμα τόκιν, Χάρι Πότερ, υπάρχει κανένας μάγος που το μπλοκάρει αυτό. μπορούμε να κάνουμε εφευρέσεις για τόσο μεγάλα και γιγαντιά έργα και δεν μπορούμε να βρούμε μια μικρή μπαταρία για ένα ηλεκτροκίνητο όχημα. Οι κακές γλώσσες λένε ότι το μπλοκάρει αυτό η βιομηχανία των ορυκτών καυσίμων. Εγώ επειδή δεν πιστεύω στα παραμύθια, ρωτάω γιατί δεν έχουμε ακόμα μπαταρίες τέτοιες. Ρωτώ τον κύριο Φέγκε, είστε του ΩΣΑ εσείς και συμμετέχουν, είπατε, πολύ περισσότερες χώρες εκεί από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Η κυρία Ντεπρέ λέει ότι βεβαίως θα πάμε πάρα πολύ καλά. Αλλά τα πάμε όντως τόσο καλά. Έχουμε την Google και όλους εκεί αυτές τις εταιρείες. Ε, ε, η Ευρώπη πώς θα πάει, γιατί έχω ακόμα την εντύπωση ότι 28 χώρες προσπαθούν όλες να εφεύρουν το αυτόματο αυτοκίνητο με βεβαίως ε, πρωτοστατούσα τη Γερμανία, αλλά όταν ε, το θέμα είναι η ουσιαστική συνεργασία, τότε δεν έχω ε, πιστεί, δεν είμαι τόσο ενθουσιώδης. Και έχω και μια ερώτηση προς την κυρία Σόφκα. Είναι μάλλον φιλοσοφική η ερώτηση αυτή, θεωρητική. Η ιδιοκτησία, κατοχή ενός γιοταχή, όταν κάποιος μένει στην πόλη, ξέρω εγώ Βαρσοβία, Ρότερνταμ, Άμστερνταμ, Βερολίνο, είναι εύκολο να έχει σύγχρονες ε, μορφές συλλογική ε, κυκλοφορίας. Αλλά όταν ζει στην Ήπεθρο και στην Ολλανδία και στην Πολωνία, το αυτοκίνητο που μπορεί να είναι ηλεκτρικό είναι ένα στοιχείο χειραφέτησης του ανθρώπου. Και ακούμε τώρα όλη μέρα εδώ ότι το ΙΟΤΑΧΗ είναι κακό πράγμα και θα το καταργήσουμε και θα πάμε όλοι σε διασυνδεδεμένα οχήματα, ηλεκτρικά, τα οποία θα μοιραζόμαστε συλλογικά. Δεν ξέρω, ξετρελαθούν οι δικοί μου εκλογείς με αυτό. Και σταματώ εδώ, Πρόεδρο. Ε, ναι, ναι, επιτρέπετε να το πεις έτσι και να κλείσει. Ναι. Ο Ισμαήλ Λερτούκ. Ευχαριστώ πολύ να Βίμ, τώρα καταλαβαίνεις γιατί μένει σε πόλη και όχι στην Ήπεθρο ο πρόεδρος μας. Κατάλαβες. Ε, μήνα, θα, το, θα τον προκαλέσει και θα αρχίσει να λέει για τα ποδήλατα, σε παρακαλώ. Καλά, την άλλη φορά. Δύο ερωτήσεις. Ε, κυρία Ντεπρέ, ε, να με χαρά να ξεκινήσω από σας. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Ε, σας άκουσα με μεγάλη προσοχή για την προστασία των δεδομένων, αλλά δεν νομίζω να ε, δίκρινα ποια είναι η άποψή σας ε, σε σχέση με την κατοχή και την ιδιοκτησία των δεδομένων. Σε ποιον ανήκουν σε τελική ανάλυση. Έχω και λόγο που το ρωτάω, πολύ συγκεκριμένο. Στην τελευταία έκθεση αυτοκινήτου στη Φραγκφούρτη ήμουνα σε ένα πάνελ και εκεί ήταν και πολλοί άλλοι ενδιαφέροντες άνθρωποι από διάφορους κλάδους τη αυτοκινητοβιομηχανίας και ανέκυψε και αυτό το ερώτημα. Ξέρω, ήταν και ασφαλιστικές εταιρείε, ε, αυτοκινητοβιομηχανίες και εγώ ίδιος ως πελάτης ενδιαφέρομαι. Και εμείς οι νομοθέτες θα πρέπει να ορίσουμε ένα πλαίσιο, αλλιώς ε, θα υπάρχουν προβλήματα. Τώρα για το πώς θα ε, προστατευτούμε από επιθέσεις hacker, αυτό το ε, θέμα δεν είναι το παρόντος, δεν θα το αναφέρω. Κύριε Φιόγκε, ε, είδαμε και ψάξαμε και βρήκαμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας στη Γερμανία έθεσε μια μελέτη στο Ινστιτούτο Fraunhofer που προτείνει να έχουμε μια προσέγγιση εξελικτική, δηλαδή όχι, όχι εξελικτική αλλά επαναστατική, δηλαδή να περάσουμε αμέσως στα αυτόματα και αυτόνομα αυτοκίνητα και να γίνει η μεγάλη κίνηση αυτή ε, στην αστική ε, κυκλοφορία. Πώς το βρίσκετε, πώς σας φαίνεται αυτό. Δηλαδή πρόσωλο ταχώς, τέρμα τα γκάζια. Αυτό είναι τεχνικά δυνατό είναι όριμο ή πρέπει να περάσουμε σε μια ήμια αυτοματοποίηση. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να έχει ζητήσει το λόγο. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός, αυτοκινητόδρομος, ε, σιδηρόδρομος σε όλη την Ευρώπη. Ε, ε, είναι υποχρεωτικό το τέλος στο σιδηρόδρομο και όχι στο αυτοκινητόδρομο. Και εδώ θέλω να επενέσω την Ελβετία. Το κατάφεραν. Δεν θέλουν να βάλουν δύο διασταγιοταχή, αλλά βάλαν στα φορτηγά πάνω από 3,5 τόνους σε όλους τους δρόμους. Δηλαδή, δεν έφυγαν από τον αυτοκινητόδρομο για να πάνε σε περιφερειακούς δρόμους, δρόμους καντονιών, ε, επαρχιακούς και τέτοια. Είχαμε πάει στην Ισπανία με την Επιτροπή με το λεωφορείο πήγαμε σε ένα νέο αυτοκινητόδρομο που χρηματοδοτήθηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε μισή ώρα περνούσε και από κάνα φορτηγό. Και μετά πήγαμε στο παλιό εθνική οθό, εκεί να δείτε φορτηγό το φορτηγό. Δηλαδή, εμείς ε, χρηματοδοτούμε μια υποδομή και δημιουργούμε έτσι το οικονομικό πλαίσιο ώστε να μην χρησιμοποιεί ψυχή. Τέτοια ηλικιότητα δεν έχει κανένα ιδιώτης. Η πολιτική πώς τα καταφέρνει. Ε, αφού έχετε το θετικό αυτό σύστημα για τα φορτηγά στην Ελβετία, εάν το μεταφέρετε και στα ΙΟΤΑΧΗ ε, δεν θα είναι καλό και ισχύει για όλους και σε όλη την επικράτεια και δεν αλλάζουν δρόμο. Και επίσης σε συγκεκριμένες ώρες της μέρας μπορεί να χρειαστεί να βάλουν και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δεν πειράζει αυτό, καλό είναι, αλλά το θέμα είναι το πρώτο να ισχύει παντού, όπως και στο σιδηρόδρομο. Και επειδή είναι και στο σιδηρόδρομο πρότυπο και παράδειγμα προ μίμηση η Ελβετία, θέλω να το δούμε αυτό. Το λόγο ζήτησε τώρα όμω ο Ντομινίκ και Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να κάνω ένα σχόλιο πρώτα. Έτσι μια γενική παρατήρηση, δεν είναι ειδική, δεν αναφέρεται στις μεταφορέ μόνο. Ότι βρισκόμαστε σε μια καμπή και γίνεται μια ρήξη εδώ. Ε, ε, εκεί που συναντάει η επιστήμη, την κοινωνία και τις συνήθειές της. Θα πρέπει ο καθένας να βρει το, το οικονομικό μοντέλο και το ρυθμιστικό. Συνήθως το οικονομικό μοντέλο έρχεται μόνο του και αυτορυθμίζεται. Η κανονική ρύθμιση νομοθεσία παίρνει περισσότερο χρόνο. Και γι' αυτό ερωτώ. Διερωτώ με δηλαδή. εκείνοι που είναι υπέρ της επανάστασης εδώ με τα αυτόνομες μεταφορές μας λένε τι, ότι θα χρειαστεί 20 χρόνια, γιατί θα χρειαστεί καιρό και η ρύθμιση. Και βλέπουμε δύο μοντέλα ε, και το είπε και ο Ισμαήλ Ερτούκ προηγουμένως ρώτησε Στην αυτόνομη οδήγηση υπάρχει ένα προοδευτικό ε, μοντέλο και ένα μοντέλο πέρ της ρήξης, δηλαδή να γίνει μεγάλη επανάσταση. Οι μεγάλες εταιρείες είναι ευρωπαϊκές και έχουν προχωρήσει σε μια προοδευτική αντικατάσταση. Η BMW προηγουμένως μας τα εξήγησε. Δηλαδή βάζουν σταδιακά χρόνο με το χρόνο νέα στοιχεία και ενοτομία στο αυτοκίνητο για να πηγαίνουμε όλο και πιο ε, κοντά σε μια αυτονομία. Όταν βάλαμε κόφτη στα αυτοκίνητα δεν έγινε και χαμός καμιά τεράστια διαβούλευση στην κοινωνία. Όταν βάλαμε λοιπόν αυτό το κόφτη που ρυθμίζει την ταχύτητα ε, δεν σημαίνει ότι ε, δεν ελέγχαμε καθόλου το αυτοκίνητο. Πήγαινε μόνο του βεβαίως κάποια στιγμή το ελέγχει αυτό το cruise control. Κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια ε, έχουμε νέες προτάσεις και εκεί δεν γίνεται ολόκληρη συζήτηση για τη ρυθμίση, την νομοθετική. Ε, και ε, για το πώς αλλάζεις σε λωρίδα, πώς ε, διασχίζεις κάποιες διαχωριστικές γραμμές, πώς κρατάς την ίδια λωρίδα όταν έχει συγκεκριμένη ταχύτητα. Όλα αυτά δεν χρειάστηκαν καμία τεράστια συζήτηση για τη ρύθμιση. Και μετά υπάρχει και το άλλο το επαναστατικό μοντέλο που είναι αυτό της Apple ή της Google που δεν λένε να έχουμε μια σταδιακή μετάβαση αλλά μια απότομη μετάβαση άρα χρειάζεται ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο και διαφορετική νομοθετική ρύθμιση. Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό κινητοβιομηχανίες που ε, σιγά σιγά ε, χτυπάνε το αυγολέμονο, ρίχνουν λίγο λίγο λίγο για να μην κόψει ε, μήπως χρειαστεί κάποια στιγμή να έχουμε συνολική αντικατάσταση. Ε, αυτό που ζητούν να γίνει τώρα και με ριζική ε, ρήξη οι εταιρείε της πληροφορικής και δεν κάνουν αυτοκινητοβιομηχανίες. Λοιπόν, μήπως έχει έρθει η ώρα οι ίδιοι οι κατασκευαστές μας στην Ευρώπη να ενδιαφερθούν για αυτό το μοντέλο της ρήξης, το επαναστατικό και όχι το εξελεκτικό. Βέβαια, το ξέρω ότι από πλευράς αγοράς αυτό είναι τεράστιο ρίσκο που θα αναλάβουν. Και Δεύτερη ερώτηση. Ποιο ε, είναι το οικονομικό μοντέλο της υποδομής, δηλαδή τώρα μιλούμε για τις φυσικές υποδομές, εντάξει ποιος χρησιμοποιεί τους δρόμους, ποιος πληρώνει ποια διόδια, τι ώρα της ημέρας, με ποια συμφόρηση, ωραία προσπαθούν οι πολιτικοί να εφεύρουν τρόπους να εισπράξουν πόρους και οι ε, καταναλωτές, οι χρήστες μάλλον των οδικών δικτύων προσπαθούν να αποφύγουν να πληρώσουν διόδια γιατί εκτιμούν ότι τα πληρώνουν απαλού. Ε, εκτός από αυτή λοιπόν την φυσική υποδομή ε, υπάρχει και μια ψηφιακή υποδομή. Το αυτοκίνητο το πληρώνει ο χρήστης. Ωραία. Αυτό είναι αυτόνομο. Είναι όμως και διασυνδεδεμένο στην αυτόματη αυτόνομη οδήγηση. Ποιος πληρώνει την ψηφιακή υποδομή και ποιο είναι το οικονομικό μοντέλο. Δηλαδή δεν θα πληρώνει διόδια. Εδώ δεν μπορούμε να εισπράξουμε διόδια για τη χρήση των δρόμων, της, της ε, φυσικής υποδομής. Την ψηφιακή ποιος θα την πληρώσει. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ερχόμαστε στις απαντήσεις. Ο κύριος Σάμψον. Νομίζω ο Μάικολ Φαραντί και ο Μεντελέγεφ φταίνε για τις ηλεκτρικές μπαταρίες, γιατί όλα είναι χημεία και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν ε, ηλεκτρογικά συστήματα τα οποία καταρχήν θα μπορούσαν να είναι πολύ μικρά, αλλά θερμαίνονται πολύ γρήγορα. Μπορεί να έχει μια μικρή λοιπόν μπαταρία, αλλά χρειάζεται ένα τεράστιο σύστημα ψήξη για να την ε, κρυώσει. Επομένω, χρειαζόμαστε διαφορετική χημεία. Κάποια στιγμή θα προκύψει, δεν ξέρω πού και πότε, αλλά είμαι βέβαιο ότι θα προκύψει. Αυτή είναι η φύση τη καινοτομία. Αν μπορούσα να κάνω ένα ε, γενικό σχόλιο για τις υπόλοιπες ερωτήσεις οι οποίες τέθησαν που ζητούν γιατί δεν κάνουμε κάτι άλλο, ιδίως όσον αφορά το οικονομικό μοντέλο. Νομίζω ότι αν βάλετε πέντε εμπειρογνώμονε σε μια αίθουσα θα πάρετε 7 διαφορετικέ απαντήσει για το γιατί πρέπει ή δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι κατά την άποψή μου ε, η λύση για να προχωρήσουμε είναι να κάνουμε δοκιμέ. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε μετολοποίηση, αλλά μπορούμε να διαπιστώσουμε. Μπορούμε να κάνουμε λογικέ δοκιμέ και θα βρούμε, με το δύσκολο μέτρο αλλά θα βρούμε. Ευχαριστώ πολύ. Για να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Ντεκάμ για τη συμμετοχή στον ΩΣΑ και τις ε, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα δω τι ε, επιδόσεις έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι είναι το γεγονός ότι σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση το Διεθνές ε, Φόρουμ Μεταφορών ζητά να μην υπάρξει ε, νομοθεσία, να κοιτάξουμε την κρυστάλλινη σφαίρα μας και να βρούμε κάποιες λύσεις. Αυτή θα ήταν η εύκολη διέξοδος. Και εμένα με ανησυχεί το θέμα αυτό. Έχω συμμετάσχει και σε προγράμματα ε, στο παρελθόν, ε, κυρίως για την αυτοματοποίηση των οχημάτων. Ε, έχω ασχοληθεί στα πρώτα προγράμματα από το 2001 το 2007. Πολλά εξ αυτών συνεχίζονται και γίνεται και πάρα πολύ καλή και συνεχίζει δουλειά από αυτών. Η πρόοδος βέβαια είναι πολύ αργή. Αυτό πρέπει να σας το ομολογήσω. Εγώ ήμουν και από το 2001 έως το 2006. Δεν ε, περίμενα να ξανασχοληθώ με το θέμα της αυτοματοποίησης των οχημάτων στην καριέρα μου, γιατί νόμιζα ότι δεν πάει πουθενά αυτή η δουλειά. Και η Google βέβαια είπε ας το δοκιμάσουμε. Μπορεί να πετάξουμε και λίγα χρήματα, αλλά όχι στην πραγματικότητα δεν πετάμε, γιατί όλο και κάτι μαθαίνουμε. Εάν υπάρχει τέτοιο πνεύμα, ίσως μπορεί να μην είχαν υποχρεωθεί οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες να ε, αναζητήσουν λίγο περισσότερα τα πράγματα. Υπάρχει το αμερικανικό μοντέλο το οποίο κυριαρχεί σε πάρα πολλούς τομείς ε, και δημιουργεί προβλήματα ίσως. Ε, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι δημιουργεί προβλήματα γιατί δεν μπορούμε να τους ακολουθήσουμε κατά πόδας. Ε, δεν ξέρω. Ακούσαμε και για τα 20 χρόνια και αλληλοεπικαλύψεις και γι' αυτά. Εγώ ανησυχώ. Ανησυχώ όταν ακούω τέτοιε δηλώσεις και νομίζω ότι πρέπει να αποφύγουμε να κάνουμε τους Ευρωπαίους ε, τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες την επόμενη Polaroid ή την επόμενη Νόκια. Φαίνεται ότι προσπαθούν ε, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και θα πρέπει να ξαναδούμε ε, από την αρχή πώς λειτουργεί η νομοθεσία και ίσως τα δεδομένα θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Η δεύτερη ερώτηση του κυρίου Έρτουχ. I have to say I haven't heard about that study and I... λοιπόν, ε, Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα. Ίσως όμως όχι στην ε, ώρα εχμής της πόλης. Ίσως θα ήταν καλή ιδέα να μην ακολουθήσουμε την παραδοσιακή οδό των αυτοκινητοβιομηχανιών να κινούμαστε με μικρά βηματάκια. Εδώ πρέπει να πούμε να το δοκιμάσουμε. Νομίζω η Σουηδία θα κάνει μεγάλα πειράματα για αυτοματοποιημένα οχήματα σε ε, διαδρομές που κάνει κάποιος για να πάει από το σπίτι του στη δουλειά του εκτός πόλεων. Ε, το συζητήσαμε αυτά. Ε, αυτοματοποιημένα φορτηγά σε αυτοκινητοδρόμους είναι ίσως ο πιο εύκολος τρόπος ε, γιατί είναι ελεγχόμενο το περιβάλλον εκεί. Τώρα, αν περάσουμε σε άλλες μορφές ε, δρόμων, αλλά όχι στις αστικές περιοχές, ε, όχι στις πόλεις, ε, υπάρχει τεχνολογία. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη νομοθεσία. Αλλά αν οι θύνοντες πούν να το δοκιμάσουμε, τότε θα το δοκιμάσουμε, θα το επιτρέψουμε από πλευρά νομοθεσία και μετά το ερώτημα το οποίο απομένει είναι αν υπάρχει κατάλληλη τεχνολογία ήδη. Νομίζω ότι για τα περισσότερα λίγο πολύ τα έχουμε. Για τα πιο μεγάλες αστικές περιοχές ε, που είναι πιο πολλές, ίσως να μην υπάρχει τεχνολογία ακόμα για να αντιμετωπίσουμε κάθε περίπτωση. Ε, μπορεί να γίνει με ασφαλή τρόπο, αλλά αυτό σημαίνει ότι σε αρκετές περιοχές θα πρέπει να είναι πολύ χαμηλή η ταχύτητα και να υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις τις οποίες το όχημα δεν θα ξέρει τι να κάνει και προκειμένου ε, να είναι ασφαλές θα μένει ακίνητο για αρκετή ώρα. Ε, θα υπάρξουν τέτοιες περιπτώσεις. Αυτές όμως είναι ακραίες περιπτώσεις. Ε, δεν σημαίνει αυτό όμως ότι ε, πρέπει να τα παρατήσουμε όλα. Ευχαριστώ, Ραφαλ Κέστη. Ευχαριστώ πολύ. Για την ερώτησή σας, κύριε Κράμερ, αν μπορούμε να έχουμε διαφοροποιημένες ε, ε, τιμολογήσεις, χρεώσεις, εμείς Ε, ορισμένοι πρέπει να πληρώσουν περισσότερα επειδή ε, είναι πιο βαρέα τα οχήματά τους και από αυτά προκύπτουν 1,5 δις τα οποία επιστρέφουν στις μεταφορές γιατί δεν έχουμε ήδη μία πολιτική τιμολόγηση που να ισχύει παντού ε, εμείς θέλουμε να την κάνουμε πολύ πιο ε, κλιμακωτή Υπάρχει και πρόβλημα αποδοχής βέβαια. Δεν είναι εύκολο να εξηγήσουμε στον πληθυσμό ότι επωφελείται και δεν υπάρχουν και πρότυπα αναφοράς που να έχουν ελεγχθεί. Για μας η καλύτερη λύση θα ήταν ακριβώς αυτή η συνολική χρέωση, αλλά νομίζω ότι δεν έχει έρθει ακόμη ώρα. Ένα σημαντικό είναι και το κόστος για να συλλέξουμε αυτά, ε, αυτές τις χρεώσεις. Βεβαίως ε, τα φορτηγά κινούνται πολύ ε, περισσότερο από τα γιοταχή. Συλλέγουμε πολλά στοιχεία για τα οχήματα, αλλά δεν τα έχουμε όλα στη διάθεσή μας, γιατί ορισμένα έχουν να κάνουν με την ιδιωτική σφαίρα. Θα μπορούσαμε να λύσουμε πολλά προβλήματα με αυτόν τον τρόπο. Ήδη την προηγούμενη Κυριακή φαίνεται ότι η κυβέρνησή μας θα συζητήσει για μια τέτοια ε, προσέγγιση του mobility pricing και θα συζητήσουμε μετά εάν θα ξεκινήσουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα και μετά θα δούμε τελικά τι ε, μοντέλο θα προτιμήσουμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η Εύα Ζόφκα. Κύριε Φαντεκάμπ, εγώ ζω στα προάστια της Βαρσοβίας και εξαρτώμαι από το ταχύ μου. Αλλά ένα ηλεκτρικό τραμ ε, ή κάτι τέτοιο θα το ήθελα. Εγώ σήμερα πηγαίνω τα παιδιά μου στο σχολείο, μετά τα πάω για ποδόσφαιρο, για μαθήματα χορού. Αλλά τι να κάνω, τέτοια γίνεται και στην Ολλανδία. Ίσως μπορούμε να το δούμε από λίγο περισσότερη απόσταση να δούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο και τα ποδήλατα, αλλά να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις πλατφόρμες ε, κυβερνοκινητικότητας για να προγραμματίσουμε τις διάφορες διαδρομές. Όταν πρέπει να πας στη δουλειά σου, δεν τηλεφωνάς στους φίλους σου. Ε, βλέπεις στο ίντερνετ ε, πότε θα ξεκινήσει ο γειτονάς σου για να πάει κάπου. Και έτσι είναι πιο πράσινη η προσέγγιση και έτσι μπορείτε ακριβώς με το γείτονά σας που θα σας πηγαίνει κάπου να γνωριστείτε και καλύτερα. Αλλά δεν είναι δυνατόν για όσους μένουν στα προάστια να εξαρτώνται αποκλειστικά από αυτά τα ηλεκτρονικά οχήματα. Ή θα πρέπει να πάρει το ποδήλατό σου ή θα εξαρτάσει από τα παραδοσιακά γιοταχήκια. Γιατί είναι τόσο διαφοροποιημένη η κατάσταση θα εξαρτασει απο τα παραδοσιακα γιοταχη γιατι ειναι τοσο διαφορετικη η κατασταση απο χωρα σε χώρα. Στην Ανδία είναι έτσι, είναι πολύ πιο όρημα κάποια συστήματα. Σε ορισμένε περιοχέ τη Ευρώπη η υποδομή δεν είναι καθόλου ε, έτοιμη για αυτοματοποίηση. Είναι άλλο θέμα εντελώ πώ θα αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κλέφντε πρέπει στο τέλο για να κλείσει. Okay. Concept of... το θέμα της ε, κυριότητας, ιδιοκτησίας, προσπαθήσαμε να το χρησιμοποιήσουμε αλλά σήμερα δεν υπάρχει κανένα νομικό κείμενο που να αντανακλά την έννοια αυτή. Θα επανέλθω στην προστασία των δεδομένων. Αυτό που υπάρχει και που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η συνένεση του ενδιαφερομένου. Όταν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, και θα επανέλθω σε αυτό, που θα, το CITS και ισχύει και για την αυτοματοποίηση, όταν παράγεις δεδομένα που μεταξύ αυτών είναι και προσωπικά, θα πρέπει ο οδηγός, του οποίου είναι τα δεδομένα, να έχει τη δυνατότητα να δίνει τη συνένεσή του ή να τον αρνείται. Αυτό ήταν και ένα τμήμα τη ε, όλη ανάλυση που κάναμε στην πλατφόρμα CITS. Ξέρετε, η έκθεση είναι αρκετά εκτενή. αλλά καταλήγει και σε κάποια λειτουργικά αποτελέσματα. Χρειάζεται ένα κουμπί που να μπορεί ε, ο, ο οδηγός να συμφωνεί να μεταδίδονται τα δεδομένα, ναι ή όχι. Ή κι άλλο κουμπί για να αποφασίζει ποια υπηρεσία θέλει και ποια όχι. Εξαρτάται κάθε φορά. Ε, μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι ε, για τις αμερικανικές σε σχέση με τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Ας μιλήσουμε ότι οι αμερικανικές εταιρείες σήμερα δεν πολλούν αυτοκίνητα ακόμα. Ακόμα. Μπορεί να βγάλουν κανένα αυτοκίνητο, αλλά ακόμα δεν πουλούν. Οπότε, εγώ δεν θέλω να είμαι εδώ εκπρόσωπος της αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά αν δεν θέλει και η αυτοκινητοβιομηχανία, πώς να το πω, να ρισκάρει τη φήμη της βγάζοντας στην αγορά αυτοκίνητα που δεν είναι 300% σίγουρα, θα έχουμε πρόβλημα. Ας μην το ξεχνάμε. Και στην Ευρώπη έχουμε μακρά παράδοση ασφαλείας. Όταν θέλουμε να έχουμε αυτή τη τεχνολογία και τις εξελίξεις, θέλουμε, αλλά για να υποστηρίζουν την ασφάλεια. Όχι για να επιδεινωθούν τα τροχιά και τα στατιστικά στοιχεία για την οδική ασφάλεια. Βεβαίω οι αμερικανικέ εταιρείε έχουν αυτή την καινοτομία, τη ρηξικέλευση με την απότομη αλλαγή. Αλλά θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ποια είναι τα επιχειρήματα της Ευρώπης υπέρ της ασφάλειας. Ευχαριστώ. Καλώ ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα ε, και συναρπαστική συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ ε, τους ομιλητές, ε, τους βουλευτές που έκαναν τις ερωτήσεις και όλους τους συμμετέχοντες. Ε, κλείνει εδώ η σημερινή μας συνεδρίαση. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Η Α, επόμενη συνεδρίαση, ξέχασα να σας πω, είναι την 5η 12 Μαΐου στις 9. Θα ψηφίσουμε για την έκθεση ΛΥΜΠΕ, τη γνωμοσοδότησή μας. Εκτάκτος, παρακαλώ, σημειώστε το. 12 Μαΐου, ημέρα 5η στις 9 το πρωί.